Αγαπητοί συνάδελφοι, να πάρουμε παρακαλώ τις θέσεις μας, διότι έχουμε ήδη καθυστερήσει την έναρξη των συνεδρία, της συνεδρίασής μας. Τελειώσαμε με καθυστέρηση, αρχίζουμε με καθυστέρηση. Σας παρακαλώ. Ο πρόεδρος Αλμπερτίνη και εγώ με τα χαρά υποδεχόμαστε τον κύριο Πουζασκάς που είναι ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκή Ένωση και ο επικεφαλής τη αντιπροσωπείας από το 2010 τη αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωση στο Αφγανιστάν μετά την έναρξη ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνα, έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα και αυτό μας φέρνει στα σημαντικά θέματα που συζητήσαμε σήμερα το πρωί σχετικά με την ΕΠΑ μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας το Αφγανιστάν είναι ένα θέατρο παράδοξο διότι από τη μια πλευρά έχουμε τα κράτη-μέλη, τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εμπλακεί από στρατιωτική άποψη, εκτός όμως από μια αποστολή, μια επιχείρηση ΕΠΑ, στα πλαίσια ενός συνασπισμού του ΝΑΤΟ που είναι παρόντα τα κράτη-μέλη μας στο Αφγανιστάν και ε, πέρα από αυτό έχουμε μια μικρή αποστολή ΕΠΑ, την ΟΠΟΛ, η οποία εστιάζεται στην κατάρτιση σε υψηλό επίπεδο της η αστυνομία του Αφγανιστάν, αλλά η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βεβαίως εκτείνεται πολύ πέρα από αυτή την αποστολή ΕΠΑ. Είναι ένας από τους σημαντικότερους παρόχους στρατιωτικής και οικονομικής και λοιπή βοήθειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει μια στρατηγική για το Πακιστάν και το Αφγανιστάν, ιδιαίτερα φιλόδοξη, τι οποίε υλοποίηση και την υλοποίηση είναι υπεύθυνο ο πρέσβη Λασφάς για τον, τον οποίο δίνω αμέσω το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων, είναι κύριε Πρόεδρε Αλμπερτίνη, με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπό την ιδιότητα ως επικεφαλής αντιπροσωπείας και της, εκπροσώπου εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Αφγανιστάν και να σας μιλήσω για τις ε, τι αντιμετωπίζει μετά τη συνθήκη της Λισαβόνα η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν. Πολλά έχουν συμβεί από τότε που σα απέφθηνα το λόγο το Μάρτιο. Τόσο από πολιτική άποψη στο Αφγανιστάν, όπου τρεις σημαντικά γεγονότα, η Τζίργα, η διάσκεψη του Καμπούλ, της Καμπούλ και οι τελευταίες εκλογές έλαβαν μέρος και σε εσωτερικό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής, της Συνθήκης Λισαβόνας που ενίσχυσαν την ΕΠΑ στην πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά από την άφηξή μου στην Καμπούλ, η αποστολή, οι δύο αποστολέ συγχωνεύτηκαν για να δημιουργήσουν την αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν αποτέλεσμα τη συνθήκη τη Αβώνα, η αντιπροσωπή ανέλαβε τι ευθύνε τη προηγούμενη αναλασσόμενη εθνική προεδρία στο Αφγανιστάν. Εγώ τώρα πλέον εκπροσωπώ, συντονίζω και διαπραγματεύομαι εξ ονόματος Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εταίρους μας του Αφγανιστάν οι επικεφαλείς των αντιπροσωπιών συναντώνται τακτικά για να αξιολογήσουν την κατάσταση στην πράξη, για να διαμορφώσουν τα πολιτικά μηνύματα και να συντονίσουν τα προγράμματα ανάπτυξης ώστε η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πιο συνεκτική και να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή το, ε, εγώ είμαι υπεύθυνο για να μεταφέρω αυτά τα μηνύματα σε όλες τις πολιτικές ομάδες, στους Αφγανούς ηγέτες και στους εκπροσώπους τη διεθνού κοινότητα του Αφγανιστάν. Με τον τρόπο αυτό προωθούμε την εφαρμογή του σχεδίου δράσης Ευρωπαϊκή Ένωση και εξασφαλίζουμε τη συνέργεια μεταξύ εξωτερική πολιτική ανάπτυξη και θεμάτων ασφαλείας του Αφγανιστάν. Η ασφάλεια των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη διεθνού κοινότητα γενικότερα είναι αρρήκτα συνδεδεμένη με την ασφάλεια και σταθερότητα του Αφγανιστάν. Είναι σαφές ότι μόνο με συντονισμένες προσπάθειες της συνολικής παγκόσμιας κοινότητας και των διεθνών οργανισμών, καθώς και άλλων πρωταγωνιστών που εμπεμβαίνουν στην πράξη, θα συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση παγκόσμιων και περιφερειακών απειλών. Τρομοκρατία, εξτρεμισμός, παράνομο, παράνομο ε, λαθρεμπόριο ναρκωτικών και οργανωμένο έγκλημα. Συνεργαζόμαστε στενά με τους συναδέλφους και φίλους, το τον, εκπρόσωπο, τον εκπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και διατηρούμε στενές σχέσεις με τον επικεφαλής του, της ISAF, τον στρατηγό Πετρέους και άλλους εκπροσώπους των διεθνών οργανισμών στο Αφγανιστάν. Παρόλο που οι εντολές μας διαφέρουν, συνεργαζόμαστε σαν ομάδα για έναν κοινό σκοπό. Ο σκοπός αυτός είναι μια μεγαλύτερη σταθερότητα στο Αφγανιστάν εντός τριών ή πέντε ετών. η κατάσταση καθίσταται πιο ασφαλής, η σταθερότητα αυξάνεται με αποτέλεσμα να μπορούμε να παραδώσουμε τις ευθύνε και τις αρμοδιότητες στους Αφγανού. ώστε να υπάρξουν αρκετά ε, εισοδήματα για να υπάρξουν βιώσιμες δομές στη χώρα που θα εξασφαλίσουν ασφάλεια και ειρήνη στο σύνολο της χώρας. Μαζί με τις ε, ε, δυνάμεις ασφαλείας του Αφγανιστάν σκοπός μας είναι να πετύχουμε όλους αυτούς τους στόχους. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης φροντίζει για την κατάρτιση των αστυνομικών και την εδραίωση του κράτους δικαίου στα πλαίσια της ευρύτερης δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει τις ικανότητες της αφγανικής κυβέρνησης αναλαμβάνοντας ορισμένες δαπάνες για την κατάρτιση αστυνομίας και για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε διάφορους τομείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης υπήρξε σημαντικός ε, στο Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη σε συνδυασμό έχουν δαπανίσει πάνω από το δισεκατομμύρια ευρώ για την ε, συνεργασία με το Αφγανιστάν. Από το 2002 συμβάλλουμε με παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο σε προγράμματα ανάπτυξης στο Αφγανιστάν και χρηματοδοτούμε του εξή τομεί. Γεωργία, αγροτική ανάπτυξη, κράτο δικαίου, διακυβέρνηση, καθώ και υγεία, τον τομέα τη υγεία. Επίση, ε, αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των δικαιωμάτων των ανδρών και των γυναικών σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Πρόσφατα υποστηρίξαμε ένα μέσο σταθερότητας στο δίκτυο γυναικών της Αφγανιστάν για την εφαρμογή των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που τονίζουν, που προωθούν τα δικαιώματα των γυναικών σε περιπτώσεις ε, κάτω από συνθήκες κρίσης και σειράξεων. Επίσης έχουμε συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη για το Αφγανιστάν. Προωθούμε τον τομέα του εμπορίου με τους γείτονες του Αφγανιστάν και προωθούμε την περιφερειακή συνεργασία μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στη, παρέχει πρόσθετα κονδύλια και υποστηρίζει την ανάπτυξη και την κατάρτιση της αστυνομίας του Αφγανιστάν. Ενισχύουμε την αγροτική ανάπτυξη, την ανάπτυξη της πέθρου και τη γεωργία, ώστε οι γεωργοί να έχουν ε, ε, βιώσιμες δυνατότητες. Ε, επίσης, χρηματοδοτούμε την ενσωμάτωση στην ε, κοινωνία των πρώην στρατιωτών οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συμβάλλουν και εκείνοι στη δημιουργία ενός ειρηνικού Αφγανιστάν. Το ΝΑΤΟ ασχολείται με το μεταβατικό σχέδιο και θα μιλήσει γι' αυτό σε λίγο ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κύριος Ρασμούνσεν. Εμείς, ως η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στοιχεία σε διάφορα επίπεδα στην Καμπούλ. Μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο για την προώθηση μεταβατικής διαδικασίας όταν ξεκινήσει μέσα της Europol με κατάρτιση στις πιο ασφαλείς επαρχίες στη φάση της, μετα... μετάβασης. Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα γεμάτη προκλήσεις η οποία έχει επηρεαστεί σημαντικά από το μακροχρόνιο πόλεμο, από τον αναλφαβητισμό και πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες ό,τι αφορά την ασφάλεια. Παρόλες αυτές τις προκλήσεις, όπως είπε, είπατε εκπρόσωπος η κυρία Άστον, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτό που υποσχέθηκε. Λαμβάνουμε μέτρα για να ευθυγραμμίσουμε τα συστήματά μας προτεραιότητες του Αφγανιστάν, να αυξήσουμε το επίπεδο της υποστήριξής μας σύμφωνα με το σχέδιο δράσης μας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως και κάποια από τα κράτη-μέλη μας συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Το 2010 χαρακτηρίζεται από μια μεγαλύτερη προθυμία τη ηγεσία του Αφγανιστάν να λάβει μεγαλύτερες ευθύνε και να οικειοποιηθεί τη διαδικασία ανάπτυξης αθερότητας της χώρας με την υποστήριξη τη διεθνού κοινότητα. Όπως αναφέρθηκε στι αρχές Ιουνίου, η Γιούργα, η οποία συγκλήθηκε, μετέφερε ένα μήνυμα Ειρηνη για συμφιλίωση και ειρήνη στο Αφγανιστάν. Πάνω από ένα πάρα πολύ υψηλό αριθμό ε, εκπροσώπων συνεδρίασαν στην Καμπούλ και χάραξαν ένα χάρτη πορεία, ένα φύλλο πορεία για συμφιλίωση και ειρήνη. Η Γιούργα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ειρήνη. Μια πλατφόρμα που μας επιτρέπει να ξεκινήσουμε ένα διάλογο με την κυβέρνηση, ώστε να υπάρξει ένας ουσιαστικός διάλογος για τη διαδικασία της συμφιλίωσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Αφγανιστάν και με τη δική μας παρότρινση και υποστήριξη 300 γυναίκες εκπροσωπήθηκαν στη Γιούργα. Αυτό εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τις οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Αφγανιστάν και συνέβαλε σε μια ευρύτερη εκτίμηση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία της χώρας. Η συμβουλευτική Γιούργα ε, συγκάλεσε ένα ειρηνευτικό συμβούλιο το οποίο όταν συσταθεί θα προγραμματίσει τη μελλοντική πορεία. Η γιούργα του, του, Ιουλίου ήταν ένα σημαντικό ορόσημο για την περαιτέρω ανάληψη ευθυνών από την κυβέρνηση του Αφγανιστάν. Ένας αριθμός αντιπροσωπιών συνήλθαν χωρίς προβλήματα ασφάλειας. Η διάσκεψη επίσης επιτυχώς πέφυγε τις παγίδες και εστιάθηκε στη διαδικασία μεταβίβασης της κυριαρχίας του Αφγανιστάν και ενίσχυσης της κυβέρνησης. Μέχρι τη διάσκεψη της Καμπούλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έπαιξε σημαντικό ρόλο εξασφαλίζοντας ότι οι υποχρώσεις από τη διάσκεψη του Λονδίνου για το κράτος δικαίου και της χρηστής διακυβέρνησης θα ενσερνίζονταν από τη νέα κυβέρνηση. Είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνή κοινότητα να εξακολουθούν να ασκούν πίεση και να πείσουν την κοινότητα να μετατρέψει τις υποχρεώσεις για χρηστή διακυβέρνηση σε απτά αποτελέσματα εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς, διότι αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Παρόλο που παρατηρούμε ότι υπάρχει ε, αποφασιστικότητα από, την πλευρά, από πλευράς, αφγανικής πλευράς να αναλάβουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις τους. Υπάρχουν διοικητικοί και δυσκολίες για την εφαρμογή αυτών των υποχρεώσεων. Ο πόλεμος έχει αφήσει τη χώρα με πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό ικανών ε, αξιωματούχων και υπαλλήλων που θα μπορούσαν να αναλάβουν ε, αποτελεσματικά το πρόγραμμα σταθερότητας και ανασυγκρότησης της χώρας. Χρειάζεται λοιπόν μία ισχυρή κυβέρνηση η οποία να στηρίζεται από τους δημοσίους υπαλλήλους Επίσης, να καταπολεμηθεί το πρόβλημα της ανεπάρκειας των δικαστηρίων, της παραβίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της εκτεταμένης διαφθοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα εστιάσει τις προσπάθειές της στα κυριότερα προβλήματα της ενίσχυσης των θεσμών και των ικανοτήτων σε πρακτικό επίπεδο και θα ζητήσει, απαιτήσει όμως δέσμευση και από την πλευρά του Αφγανιστάν για την προώθηση όλων των απαιτουμένων μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς. Μετά από αίτημα των ηγετών του Αφγανιστάν πρόσφατα άρχισε να αντιλευνώ τη δυνατότητα μια συντονισμένη υποστήριξη από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων μέσω ενός δικτύου περιφερειακών κέντρων κατάρτισης στην Καμπούλ και σε άλλες περιοχές. Θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε την κατάρτιση των υπαλλήλων του Αφγανιστάν σε όλους τους τομείς και ειδικότερα στον τομέα της δικαιοσύνης. Όπως όλοι γνωρίζετε, στις 18 Σεπτεμβρίου οι πρώτες κοινοβουλευτικές βουλευτικές εκλογές έγιναν μετά από το 2001. Παρόλο που είναι ακόμα πάρα πολύ νωρί να πούμε οτιδήποτε για τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών, ε, αποτελούν ε, μια σαφή ένδειξη υποστήριξη τη κυριαρχία του Αφγανιστάν. Ολοκληρώθηκαν κάτω από δύσκολε συνθήκε οι εκλογέ αυτέ. Το ότι η διεξαγωγή εκλογών κάτω από αυτέ τι συνθήκε μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα επίτευγμα από μόνο του. Εγώ πήγα στα εκλογικά κέντρα στην Καμπούλ και πραγματικά εντυπωσιάστηκα και συγκινήθηκα από το θάρρος του λαού του Αφγανιστάν που άσκησε τα δημοκρατικά του δικαιώματα παρόλο το δύσκολο περιβάλλον ασφαλείας, τον εκφοβισμό και τις απειλές. 4,3 ψήφοι ε, συγκεντρώθηκαν, 30 40% του εκλογικού σώματος. Σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές σημειώσαμε καλύτερη οργάνωση με αποτέλεσμα να ανακοινωθούν τα εκλογικά κέντρα ένα μήνα νωρίτερα που είναι σημαντική βελτίωση σε σχέση με αυτά που είχαν συμβεί το 2009 όταν ανακοινώθηκαν τα εκλογικά κέντρα δύο μέρες μόλις πριν από τις εκλογές σημείωσα ότι υπήρχε μεγαλύτερη διαφάνεια και, πιο, και μια διαδικασία λήψη αποφάσεων πολύ πιο ουσιαστική και διαφανής. Οι αποφάσεις ε, που είχαν ληφθεί για, να λειτουργήσουν, για να λειτουργήσουν όλα τα εκλογικά κέντρα τηρήθηκαν παρόλο που είχαν ε, ε, ασκηθεί πιέσεις για να αυξηθεί ο αριθμός των εκλογικών κέντρων. Επίσης υπήρξε μεγάλος αριθμός ε, νέων και γυναικών που ήταν υποψήφοι στις εκλογές. Υποστηρίζουμε, είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε αυτούς τους θαραλέους νέους και τις θαραλέες γυναίκες τους επόμενους μήνες. Αλλά οι εκλογές δεν είναι το παν. Μπορεί τα αποτελέσματα να ήταν γενικά ικανοποιητικά αλλά οφείλεται αυτό το αποτέλεσμα και χάρη στην σημαντική υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας των Ηνωμένων Εθνών και στις προσπάθειες των δυναμέων ασφαλείας ε, του Αφγανιστάν. Παρ' όλα τα αυτά όμως η περίοδος τώρα είναι κρίσιμη καθώς γίνεται επεξεργασία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Κάτι που θα συνεχιστεί για ένα διάστημα και κάτι που θα οδηγήσει σε τεχνικές και πολιτικές προκλήσεις. Προκαταρκτικά αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να ανακοινώνονται από διάφορες επαρχίες. Υπήρξε οπωσδήποτε καλπονοθεία. Είναι η αρμόδια, αμφισβητείται η, αρμόδια, η αρμοδιότητα των εκλογικών, των εφορευτικών επιτροπών. Αλλά καθώς συνεχίζεται η διαδικασία επεξεργασίας των αποτελεσμάτων πρέπει να υποστηρίξουμε εκείνους που θέλουν να ανακοινώσουν τελικά αξιόπιστα αποτελέσματα. Πρέπει ως Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσουμε τις προσπάθειες οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει τα αποτελέσματα των εκλογών δεν είναι κάτι που εμείς μπορούμε να θεωρούμε ως ελεύθερες ε, ανεξάρτητες εκλογές. Αυτό που χρειάζεται είναι να εξασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα θα γίνει αποδεκτό. Αυτές οι εκλογές κατά την άποψή μου εκδηλώνουν τη βούληση του λαού του Αφγανιστάν να διαμορφώσει το μέλλον της χώρας του και, το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί είμαστε στο Αφγανιστάν παρόντες για να εξασφαλίσουμε την, την μελλοντική ανάπτυξη, ασφάλεια και ευημερία αυτή, αυτής της χώρας. Γίνονται προσπάθειες για τη σταθεροποίηση του Αφγανιστάν με 250 μέλη προσωπικού από 23 κράτη-μέλη καταβάλουμε προσπάθειες για την αστυνόμευση και για την ασφάλεια της χώρας. Εγώ έχω εντολή να παρέχω στη Europol την, πολιτική, την απαιτούμενη πολιτική καθοδήγηση. Επισκέπτομαι με εκπροσώπους της Europol τις διάφορες επαρχίες, ενημερώνω για τις δραστηριότητες με τον, είμαι, με τον, έχω πολύ στενή σχέση και συνεργασία με τον επικεφαλή τη Γιουπόλ όπω και με τον προηγούμενο. Και τώρα μου δόθηκε μια ευκαιρία να σα ενημερώσω για αυτά τα οποία έχουν συμβεί και να ανταλλάξω μαζί σα ορισμένε απόψει για το τι θα μπορούσε να γίνει από εδώ και πέρα. Όπως ξέρετε υπάρχουν έξι στρατηγικοί ε, στόχοι που σχετίζονται με τις ικανότητες της UPOL έτσι ώστε να ενταχθούν σε ένα λειτουργικό πλαίσιο. Καταρχήν έλεγχος της αστυνομίας, υπηρεσία πληροφοριών και ένα τμήμα εγκληματολογίας στο Υπουργείο Εξωτερικών καταπολέμηση της διαφθοράς, συνεργασία δικαιοσύνης και αστυνομίας και επίσης σύσταση τμήματος προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης υπάρχει ένα πρόβλημα για την συγκρότηση της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. 125 ε, μαθήματα χορηγήθηκαν σε 11.000 αστυνομικούς. Η Ιούπολ επίσης ε, προέταξε 260 σχέδια μέσα στα πλαίσια ε, ενός σχεδίου λειτουργίας και μεταρρύθμισης των αστυνομικών δυνάμεων. Άρα έγινε κατάρτιση 15.000 ωρών έτσι ώστε αυτά τα σχέδια κατάρτιση να ενταχθούν. Επίσης η UPOL ήθελε να καταπολεμήσει τη διαφθορά και όπως ξέρετε υπάρχει τμήμα καταπολέμησης της διαφθοράς ε, μαζί με την MOI και την Εθνική Αστυνομία. Θα πρέπει όμως να δούμε την ευρύτερη εικόνα και να αναγνωρίσουμε ότι η υπηρεσία κατάρτισης του ΝΑΤΟ και η σύστικα ε, των ΙΠΑ είναι η βασική εμπλεκόμενη φορείς για την ε, κατάρτιση και για τη μεταρρύθμιση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Επίσης, το ΝΑΤΟ συνεισφέρει και μπορεί να χρησιμοποιήσει συμβαλόμενο ε, συμβασιούχους έτσι ώστε να ε, εφαρμόσουν αυτό το σχέδιο. Υπάρχει ένας ε, επιχειρησιακός προϋπολογισμός που είναι πολύ υψηλός ενώ μόνο 58 εκατομμύρια αφορούν το κοινοτικό προϋπολογισμό. Ενώ λοιπόν υπάρχει συνεργασία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Καμπούλ, Βλέπουμε ότι υπάρχει περιθωριοποίηση αυτή της υπηρεσίας μέσα στα πλαίσια των μεταρρυθμίσεων εάν δεν δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό το τομέα. Τα κράτη-μέλη και το Αφγανιστάν θεωρούν ότι η UPOL δεν εστιάζει την προσοχή της εκεί που θα έπρεπε και θα έπρεπε να δώσει πιο χειροπιαστά αποτελέσματα. Η UPOL λοιπόν θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή σε συγκεκριμένους τομείς σε τομείς δηλαδή όπου μπορεί να χορηγήσει προστιθέμενη αξία. Θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη ικανοτήτων για τις αστυνομικές δυνάμεις και η UPOL θα πρέπει να προωθήσει και τις υπηρεσίες χωροφυλακής. Πιστεύω ότι η UPOL μπορεί να το αναπτύξει αυτό. Θα πρέπει λοιπόν η UPOL να έχει τους κατάλληλους πόρους για την εκπαίδευση και κατάρτιση σε ευρύτερη κλίμακα. Επίσης, η διμερής χρηματοδότηση δεν απέδωσε όσο θα έπρεπε για μαθήματα κατάρτισης. Δόθηκαν 500.000 ευρώ για το 2010 που είναι αμεληταία ποσότητα. Γι' αυτό η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χορηγήσει 15 εκατομμύρια ευρώ μέσα στα πλαίσια του μέσου σταθερότητος και των περιφερειακών ε, κέντρων λειτουργίας της αστυνομίας όπου τα κέντρα αυτά θα επιτηρεί η Γιούπολ. Η Ιούπολ θα είναι η πρώτη δύναμη η οποία θα μπορέσει να καταρτήσει αυτές τις υπηρεσίες αστυνομίας και χωροφυλακής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης θα πρέπει να δώσει επιπρόσθετη υποστήριξη μέσα στα πλαίσια του μέσου συνεργασίας και ανάπτυξης. Άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, επιδοτήσουν τη UPOL έτσι ώστε να μπορέσει να προβάλλει αυτές τις ε, πολιτικές ικανότητες, δηλαδή στο τομέα της αστυνομίας και της δικαιοσύνης. Να υποστηρίξουμε μέσω προσωπικού και να μπορέσουμε να έχουμε νέους συμβασιούχους χρησιμοποιώντας και αυτούς και τους αστυνομικούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί πρόσφατα. Έτσι θα μπορέσουμε να προωθήσουμε αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις χωροφυλακής μέσα στα πλαίσια της ΕΠΑ. Κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να επικεντρωθεί σε ορισμένες εθνικές προτεραιότητες στο Αφγανιστάν. Θα πρέπει να αυξήσουμε την παρουσία μας και να προβάλλουμε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση μέσα στα πλαίσια των, κοινων, των ε, κοινοτικών αξιών, ενώ ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μία μείωση ως προς τις ε, στρατιωτικές δαπάνες στο μέλλον. Υπάρχει άμεση συνδεσιμότητα με θέματα ασφαλείας, γι' αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι εκλογές δεν είναι μόνο ένα ορόσημο είναι ένα εφαλτήριο έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει το ρόλο που της αρμόζει και ελπίζω να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα μακρόπνο σχέδιο, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να ορίσουμε τα διεθνή προγράμματα έτσι ώστε να προωθήσουμε την περιφερειακή οικονομική συνεργασία και με τις γείτονες χώρες του Αφγανιστάν. Επίσης, στα πλαίσια της ΕΠΑ θα πρέπει να προωθηθούν όλες αυτές οι συνιστώσεις και θα συνεργαστούμε και με το ΝΑΤΟ, με τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους φορείς για να προωθήσουμε αυτούς τους στόχους τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακολουθούν οι βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν θυμίζω ότι μπορούν βεβαίως να συμμετέχουν και οι εθνικοί βουλευτές ζητήστε το λόγο εάν θέλετε να μιλήσετε και βεβαίως έχετε δικαίωμα επειδή όμως έχουμε χρονικούς περιορισμούς και με την πρωινή εμπειρία θα είμαι πάρα πολύ αυστηρός ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θα έρθει στις 4 ώρα ακριβώς Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω να είστε σχετικά σύντομοι στα σχόλια και τις ερωτήσεις σας για να μπορέσουμε να έχουμε συζήτηση επί της ουσίας. Αλλά να τελειώσουμε στην ώρα μας. Ο κύριος Αρλάκη που είναι εισηγητής μας για το Αφγανιστάν. Παρακαλώ. Thank you. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστώ εξοχότατε για την ε, περιγραφή της ε, κατάστασης και τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Λίγους μήνες μόνο έχετε εκεί από αφού αναλάβατε καθήκοντα, οπότε δεν θα ήταν και δίκαιο να σας ε, ρωτήσουμε πάρα πολλά, να απαιτούμε από σας πολλά. Είναι περίπλοκη χώρα και εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Εγώ θα προτιμούσα όμως, για να το πω ειλικρινά, μια πιο ρεαλιστική περιγραφή της κατάσταση στο Αφγανιστάν και της επιρροή τη Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Γιατί μας τα λέτε ρόδινα. Και αυτό λίγο με ανησυχεί έτσι ως τοποθέτηση. Σχεδόν δεν αναφέρατε ότι εδώ και 9 χρόνια είναι σε εμπόλεμη κατάσταση το Αφγανιστάν και ό,τι και να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον πολιτικό τομέα με την αποστολή, τη Γιούπολ και τα λοιπά, ωραία, της διεθνούς ε, συνεργασίας και βοήθειας, ε, δεν μπορούν να παραγνωρίσουν αυτό το γεγονός. Ότι ό,τι και να κάνουμε εμείς, ο πόλεμος συνεχίζεται. Και υπάρχει στενή σχέση. Μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει στρατηγική. Το πρόγραμμα δράσης είναι εξαιρετικά ε, αδύναμο. Είναι ένα ευχολόγιο καλές οι προθέσεις, δεν λέω. Αλλά δεν υπάρχει στρατηγική γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ αυτών που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και του πολέμου χωρίς νικητή που σοβεί εκεί 9 χρόνια. Η ερευνητική διαδικασία είναι στα σπάρανα και θα πρέπει να πει κάτι πιο σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ειρηνευτική προσπάθεια πολιτικά και πώς συνδέεται αυτό με τη φτώχεια και τη διαφθορά που δεν φαίνεται να μειώνονται. Είναι από τις πιο φτωχές χώρες στο Αφγανιστάν του κόσμου και μετά από 9 χρόνια μεγάλης ε, παρέμβασης και βοήθειας διεθνούς. Και το θέμα της βίας. Ε, χάνουν τη ζωή τους άμαχοι. Και αυτό ανησυχεί και την αφγανική κυβέρνηση και τη διεθνή κοινότητα. Θα προτιμούσα λοιπόν μια πιο ρεαλιστική και προσεκτική περιγραφή της κατάστασης. Μου άρεσε πολύ η περιγραφή που κάνατε για τη Ιούπολ και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον συνειδητοποιεί με τρόπο πιο ρεαλιστικό το τι μπορεί να κάνει η Ιούπολ στο Αφγανιστάν. Και το θέμα ε, της ε, συνεργασίας με ε, την εκπαίδευση του ΝΑΤΟ που είναι πολύ σημαντική είναι μια καλή προσπάθεια για να ε, ε, δημιουργηθεί αστυνομία. Και πρέπει να πω ότι η χρηματοδότηση της Γιούπολο χρειάζεται σε σχέση με τα κύρια που δαπανούν οι Αμερικανοί για τη στρατιωτική εκπαίδευση. Και η Γιούπολ δεν θα πρέπει να περιθωροποιηθεί αλλά να ενταχθεί στο βασικό κορμό της διεθνούς δράσης για να μπορέσει το Αφγανιστάν να είναι ελεύθερο ξένων ε, επεμβάσεων σε τρία-τέσσερα χρόνια. Τώρα το Κοινοβούλιο συζητάει μια στρατηγική, ελπίζω σε λίγου μήνε να την έχουμε διαρθρώσει καλύτερα και να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε στο Αφγανιστάν ω Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να συνεργαστούμε στενότερα και με εσά ε, και με τι υπηρεσίε. Πάντω αξίζεται την υποστήριξή μα και σα εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Merci. La parole... Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπέρμαν που είναι πρόεδρος της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αφγανιστάν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στα αγγλικά, κύριο Σπέρμαν. Ευχαριστώ, ε, αγαπητέ Ουσέσκα. Έχω τέσσερις ερωτήσεις και δεν θα φιλολογήσω συγκεκριμένε ερωτήσεις. Κατά την άποψή σα, ποια είναι η αξία εκλογών χωρίς εκλογικούς καταλόγους, χωρίς ένα κατάλογο όπου κάθε ψηφοφόρο να έχει το όνομά του και να συνδέεται με ένα εκλογικό τμήμα. τι άλλη αξία έχουν παρά να αυξηθεί ακόμα η απαξίωση των θεσμών των ίδιων που χρειάζεται το Αφγανιστάν. Στη συνέχεια, ερώτηση δεύτερη. Χρειάζονται ενίσχυση αυτοί οι οργανισμοί και οι θεσμοί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεργαστεί βεβαίως. Θα έρθουμε σε επαφή με τη Ζήργα και εμείς και να θα δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το τοπικό κοινοβούλιο στην Καμπούλ. Όλα αυτά καλά και ωραία θα έπρεπε να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με εκπλήσει ε, που το αναφέρετε, γιατί επίσημα εδώ και χρόνια είναι αυτή η αποστολή μας. Και κανονικά θα έπρεπε να είμαστε ηγέτες σε αυτό το τομέα και να εκπαιδεύουμε νέες γενιές δημοσίων υπαλλήλων. Τι πρέπει να κάνει και τι μπορεί να κάνει καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, Τρίτον, τη UPOL. Πολύ ωραίο είναι το πρόγραμμα, το έργο δυσκολίες αντιμετωπίζει όμως, για να το πω έτσι, και θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή. Είτε θα συνεχίσουμε είτε θα σταματήσουμε. Συνέχεια σημαίνει όμως και επένδυση και σημαίνει καλύτερη εστίαση σε εκπαίδευση αστυνομικών, πολιτική και τίποτα άλλο. Ούτε στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ είναι στρατιωτική οργάνωση, στρατιωτικός οργανισμός και η αστική εκπαίδευση αστυνομικών δεν είναι θέμα των στρατιωτικών. Το αντίθετο. Είναι θέμα πολιτικό και όχι στην ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η άποψή μου και θα το συζητήσουμε με τον κύριο Αρλάκη στις τροπολογίες της έκθεσής του. Εσείς λοιπόν πώς το βλέπετε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιούπολ πώς πρέπει να εστιάζεται και πού. Το τέταρτο που δεν αναφέρεται μέχρι τώρα τόσο πολύ είναι η διαφθορά η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι ε, δωρητές υπονομεύουν νομίζω την ανάπτυξη του Αφγανιστάν δεχόμενη μια πολύ υψηλή ε, διαφθορά και ε, δωροδοκία. Και στην Καμπούλ, στη Σύνοδο Κορυφής, ο ίδιος Καρζάη καμιά φορά σταματάει τις έρευνες για διεφθαρμένους υπαλλήλους μόλις φτάνει στο περιβάλλον του αυτή η έρευνα και δεν λέμε τίποτα. Και μετά ξέρω ότι ε, είναι πλήρως εξαρτημένο το Αφγανιστάν από την ξένη βοήθεια, αλλά κάπου δεν θα πρέπει να βάλουμε και όρους. Ε, είναι αναπόφευκτο. Πώς το σχολιάζετε αυτό και τι συνιστάτε. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολλοί ομιλητέ που έχουν ζητήσει το λόγο. Θα σα παρακαλέσω να περιοριστείτε σε δύο λεπτά έκαστο. Μία ερώτηση, ένα σχόλιο, το πολύ πολύ αν γίνεται. Δύο λεπτά έκαστο. Ο κύριο Ζιγκέρη πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Λιθουανικής Βουλής. Uh, ε, αγαπητέ πρέσβη, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για τη συνεισφορά σας αυτές τις ε, δύσκολες στιγμές και σε αυτό τον κέριο τόπο για μας. Θυμόσαστε ότι οι Λιθουανοί, εμείς οι Λιθουανοί είμαστε βασικοί διαπραγματευτές και θυμόσαστε ότι και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων προσχώρησης είχαμε να αντιμετωπίσουμε πολλά θέματα ιδεολογίας ως προς την ε, κοινωνία των πολιτών. Δεν ξέρω κατά πόσο θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε υπέρ ή κατά της κοινωνίας των πολιτών. Έχουμε μια μεγάλη κληρονομιά. Οι ιδέες του Τζέφερσον και της Γαλλικής Επανάστασης βρίσκονται πολύ μακριά από την αφγανική πραγματικότητα. Πώς μπορείτε να εφαρμόσετε εκπαιδευτικά προγράμματα τη στιγμή που υπάρχουν διαφορετικά σχολεία για αγόρια και διαφορετικά για κορίτσια. Πώς θα υπάρχει λαϊκή εκπαίδευση, κοσμική εκπαίδευση σε μια χώρα η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από τις ευρωπαϊκές αξίες. Πώς θα πληρωθεί αυτό το χάσμα και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία των πολιτών, το πολιτικό σκέλος γενικά, που δεν σχετίζεται με τις ε, στρατιωτικές νίκες, αλλά αφορά τις ιδεολογικές νίκες. Η πολιτική γειτονία και στο Μεσανατολικό αφορά θέματα θρησκευτικού χαρακτήρα. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει το κοσμικό σκέλος. Εδώ μιλάτε για μία περιοχή η οποία βρίσκεται πολύ μακριά από την Ευρώπη. Δεν μπορούμε να προωθήσουμε σχέσεις γειτονίας. Πώς μπορεί να πληρωθεί αυτό το χάσμα μεταξύ ημών και της αφγανικής κοινωνίας. Η κυρία Κοπά. Thank you. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, χρησιμοποιήσατε διπλωματική γλώσσα σε σχέση με τις εκλογές στο Αφγανιστάν και δεν ξέρω κατά πόσο κατανόησα απόλυτα αυτά που είπατε. Μιλήσατε για διτά κριτήρια. Δηλαδή υπάρχουν ευρωπαϊκά κριτήρια για την Ευρώπη και υπάρχουν ε, κριτήρια τα οποία είναι καλά για τους τριτοκοσμητικούς, για να το πούμε έτσι. Μπορείτε να μας το επιβεβαιώσετε αυτό. Όλοι ξέρουμε ότι υπήρξε βία και ενωθεία το Reuters λέει ότι τουλάχιστον 17 σκοτώθηκαν σε επιθέσεις ανά τη χώρα. Επίσης, η Επιτροπή Δίκαιων Εκλογών, η Επιτροπή Εποπτείας είδαν ότι δυστυχώς έγινε μεγάλη νοθεία στις περισσότερες περιφέρειες. Δυστυχώς η όλη διαδικασία αντί να ενισχύσει την νομιμότητα του πολιτικού συστήματος μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη καχυποψία κατά, που να ταχθεί κατά της διεθνούς παρέμβασης. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τοπικούς αρχηγούς και φυλάρχους. Γι' αυτό νομίζω ότι εμείς ως διεθνής κοινότητα δεν χρησιμοποιήσαμε την προγενέστερη πείρα μας στο Αφγανιστάν όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βόλτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Απλή ερώτησή μου να ευχαριστήσω καταρχήν τον πρέσβη για την παρουσίαση και γιατί μας ε, μίλησε για μία άκρος απογοητευτική δουλειά. Το 90% της ηρωίνης στους δρόμους της Ευρώπης προέρχεται από το Αφγανιστάν. Και το κόστος τους εθνικούς προϋπολογισμούς πολέμησης της εγκληματικότητας ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια. Επίσης, η χρηματοδότηση των ανταρτών σχετίζεται με αυτό το εμπόριο, άμεσα με αυτό το εμπόριο ναρκωτικών. Όπως ξέρετε, οι περιφέρειες ε, σχετίζονται με την καλλιέργεια, άρα η εκρίζωση αυτών των καλλιεργειών θα οδηγούσε σε φτώχεια. Τα Ηνωμένα Έθνη θεωρούν ότι το κέρδος είναι της τάξης του ενός δις δολάρια ετησίως. Αυτό είναι ψυχία σε σχέση με τα χρηματικά μέσα που διαθέτουν η ΕΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βοήθεια. Δηλαδή αγοράζουμε καλλιέργειες που κανένας δεν θέλει και μετά τις αποθηκεύουμε μέχρι ότου τις πετάξουμε. Γιατί να μην αγοράσουμε λοιπόν όπιο, παπαρούνα δηλαδή, και μετά οι γεωργοί, οι αγρότες να ελέγχουν την ποιότητα. Δηλαδή να υπάρχει μία σχέση εξάρτησης, αλλά εδώ μιλάμε για ουσιώδη εξάρτηση. Επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε μία ε, πραγματογνωμοσύνη δευτέρου ε, βαθμού της τάξης του set aside. Δηλαδή μπορούμε να πληρώσουμε τους γεωργούς για το έτος συν 3, συν 4, συν 5 για να καλλιεργήσουν εναλλακτικέ ε, καλλιέργειες και να έχουν εναλλακτική συγκομιδή. Αν λοιπόν καλλιεργήσουν εκ νέου παπαρούνα, τότε μπορούμε να καταστρέψουμε την παραγωγή. Κύριε Πρέσβη, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε το εξής δεν θα πρέπει να υπάρχει μια ε, πιο ριζοσπαστική προσέγγιση γιατί η χρηματοδότηση ε, του Αντάρτικου είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να απασχολεί στην ευρωπαϊκή κοινότητα στο μέλλον. Η κυρία Άννα Γκόμες και μετά ο πρέσβης. Κύριε πρέσβη, δεν συμμερίζομαι αυτά που μας είπατε ως προς την, ε, τις εκτιμήσεις δηλαδή κατά πόσο μπορούν να ε, αποτιμηθούν οι εκλογές ως ελεύθερες και δίκαιες. Όπως είπε και η κυρία Κοπά, δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε τον πύχη σε σχέση με τις εκλογές του Αφγανιστάν. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικά κριτήρια αποτίμησης. Μιλάμε για μαζική νοθεία και βία πέρα από τις ε, συνθήκες ασφαλείας που αποτέλεσαν τροχοπέδι για πολλούς ανθρώπους. Δεν μπόρεσαν να μεταβούν δηλαδή και να ε, ψηφίσουν ως προς τη Γιούπολ. Γιατί δεν έχουμε την σωστή προσέγγιση ε, ως προς την κατάρτιση της αστυνομίας του Αφγανιστάν ως προς την ε, τάξη δικαίου θα ήθελα να πω τι ισχύει στον τομέα της δικαιοσύνης. Δηλαδή, έχει νόημα να καταρτίζετε τους αστυνομικούς τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτόνομη δικαιοσύνη, η οποία στην ουσία υποθάλπει την βία και την οθεία. Ποιο είναι το σχέδιό σας ως προς τις σχέσεις Αφγανιστάν-Πακιστάν. Ποιες είναι οι σχέσεις σας με τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στο Πακιστάν και τέλος, είπατε στους εκπροσώπους τον είπα, ότι το, όταν, ότι, το χρησιμοποιούν μη επανδρομένα εμ, μη επανδρομένα αεροπλάνα θα μπορεί να ήταν κάτι απόλυτα καταστροφικό στα, στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Κύριε Πρέσβη, ε, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Yes, uh, Επτά λεπτά. Μάλιστα. Δέκα λεπτά ήταν οι ερωτήσεις, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα καταρχάς να πω σε όλους ότι πολύ σκληρές ερωτήσεις μου κάνετε και ενδιαφέρουσες και ευχαριστώ γι' αυτό. Γιατί έτσι θα με βοηθήσει αυτό να δώσω τα μηνύματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών στο Αφγανιστάν. Το είπα και στον πρόεδρο Καρζάη πριν έρθω στις Βρυξέλλες. Ότι θα με σουβλήσουν, θα με πιέσουν, θα μου κάνουν σκληρές και δύσκολες ερωτήσεις στο Κοινοβούλιο. Και ο κύριος Σαρολάκη και πολλοί άλλοι βουλευτές ε, αναφέρθηκαν στη συμπεριφορά μου και στη στάση μου ότι τα λέω πολύ ρόδινα και πολύ αισιόδοξα. Μα είναι τόσο θολό το τοπίο, αν δεν είσαι αισιόδοξο, ζωφερό το τοπίο, αν δεν είσαι αισιόδοξο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είμαστε λοιπόν συγκρατημένα αισιόδοξοι, αλλιώ δεν θα δουλεύαμε. Καταλαβαίνω αυτά που λέτε και τις παραμέτρους. Βεβαίως και έχουμε τα ίδια κριτήρια και θέλουμε να έχουμε τα ίδια κριτήρια, κυρία Γκόμες, και για τους Αφγανούς. Και θέλουμε να δούμε τις ίδιες εκλογές, όπως και στη Λιθουανία και την Ελβετία. Αλλά δεν είναι του παρόντος αυτό, ούτε αύριο θα γίνει. Και θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και στους ε, αξιότιμους φορολογουμένους στο θεωρείο. Γιατί δεν είναι χώρα που ζούσε 9 χρόνια πόλεμο. 30 χρόνια είχε εσωτερικές σειράξεις και πάει λέγοντας. 80% του κόσμου είναι αγράμματοι, είναι αναλφάβητοι. Πρόκειται για μια χώρα που δεν γνωρίζει ούτε ο πρόεδρος Καρζάη, ούτε ο στρατηγός Πετρέους, ούτε ο κύριος Ομπάμα πόσοι είναι οι κάτοικοι της χώρας. Πόσους Αφγανούς έχει το Αφγανιστάν. Να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν λέω ε, να κάνουν την εκλογική μεταρρύθμιση αμέσως μετά τον Οκτώβριο, αλλά και για τον εκλογικό κατάλογο. Είναι κρίσιμο βεβαίως και προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε δημοκρατική εκλογική αναμέτρηση. Και θα πρέπει να έχουμε το σθένος να γίνει η μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου και ε, με την έννοια της μίας ψήφου που να μην μεταβιβάζεται που, γιατί ε, είναι μεγάλο εμπόδιο αυτή τη στιγμή αυτό που ισχύει για την ανάπτυξη πολιτικών κινημάτων και κομμάτων στο Αφγανιστάν. Οπότε η απάντησή είναι βεβαίω είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι σκληρή. Οι εκλογέ ε, είχαν και βία τη μέρα των εκλογών. Πώ να μην υποστηρίξουμε ένα λαό που παρά αυτέ τι απειλέ και αυτή τη βία πήγε και ψήφισε, πήγε στι κάλπε. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη ενθάρρυνση που έχω ζήσει τις τελευταίους έξι μήνες στο Αφγανιστάν. Αν μου επιτρέπετε να επανέλθω σε πιο ειδικέ ερωτήσεις που έγιναν. Ο κύριος Αρλάκη και πάλι. Σας ευχαριστώ και εκτιμώ το ενδιαφέρον σα και ε, παρακολουθώ και τις συζητήσεις, το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά κατά την ταπεινή μου άποψη, στρατηγική έχουμε. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να σκουμποθούμε και να δουλέψουμε ε, επιτόπου με υποστήριξή σας για όλες τις ε, ε, μεταρρυθμίσεις και για την αύξηση του δυναμικού της Γιούπολ γιατί χρειάζεται βοήθεια από τα κράτη-μέλη. Βοηθήστε μας σας παρακαλούμε. Και στη συνέχεια ο Τάις Μπέρμαν με ρώτησε διάφορα πράγματα. Τι πιστεύετε για τους εκλογικούς καταλόγους σας απάντησα. Για τους θεσμούς και πάλι αυτό είναι κατοχυρωμένο στο πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια εμπειρία για το πώς λειτουργεί εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το μαρτυρά και η δική μου παρουσία εδώ ενώπιόν σας. Κάνουμε ε, ε, προγράμματα για την ανάπτυξη ας πούμε και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι πολλές οι προκλήσεις για το Αφγανιστάν. Στο UNDP έχουμε ταχύρυθμα ας πούμε, ε, τμήματα, πενθήμερα για την εκπαίδευση και σεμινάρια, η διαδικασία λήψη αποφάσεων, η διαβουλεύσεων ε, μεταξύ των διαφόρων φορέων και οργανισμών. Ε, Βεβαίω παραμένουν ακόμα πολλά να γίνουν για να υπάρχουν απλοί οργανισμοί και ξέρω ότι οι Γάλλοι, οι Βρετανοί θα μας βοηθήσουν και οι Σλοβαίνοι τώρα για τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών. και ε, χρειάζονται ε, κέντρα εκπαίδευσης, δημόσια δίκησης για τη μελλοντική ε, ελίτ που θα είναι οι νέοι ηγέτες του Αφγανιστάν. Και ελπίζω να μας υποστηρίξετε και εκεί καθώς προχωρούμε σε αυτή την προσπάθεια που δημιουργούμε σχολές και, για τη δημόσια διοίκηση στη χώρα. Στη συνέχεια, για τη Γιούπολ. Βεβαίως. Έξι είναι οι στρατηγικοί στόχοι και πάλι οι στόχοι αυτοί αντανακλούν την πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ήταν προϊόν συμβιβασμών και συνένεσης μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Ο κόσμος εκεί είναι πολύ αφουσιωμένος και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και σημαντική. Αλλά έχουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Όπως είπε και ο κύριος Σαρλάκη, θα παρακαλούσα και εγώ να επικεντρωθούμε σε μία προτεραιότητα. Και αυτό το αναγνωρίζουν και οι Αφγανοί και οι φίλοι μας οι Αμερικανοί τώρα που έρχονται με πολλά χρήματα. Αλλά κανένας δεν έχει τη δυνατότητα και την εμπειρία της Γιούπολ που είναι η εκπαίδευση, η πολιτική εκπαίδευση αστυνομικών. Και πρέπει να διοχετεύσουμε εκεί, πιστεύω, περισσότερους πόρους για να κάνουμε μια πολύ ε, σκόπιμη επένδυση. Όχι να εκπαιδεύουμε παραστρατιωτική αστυνομία, γιατί αυτό τώρα γίνεται, γιατί όντως χρειάζεται, αλλά ναι, είναι πραγματική πολιτική αστυνομία και να λογοδοτεί. Και μια τελευταία ερώτηση που κάνατε κι εσείς και άλλοι είναι η διαφθορά. Βεβαίως, μεγάλο ζήτημα αυτό. Γι' αυτό εγώ ηγούμε των προσπαθειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξ ονόματος της διεθνούς κοινότητας για να αντιμετωπιστεί πριν από τη διάσκεψη της Καμπούλ. Ε, χαίρομαι που βρήκε και τη θέση του στη ε, δήλωση της Καμπούλ, αλλά τώρα θα πρέπει οι δηλώσεις προθέσεων να γίνουν αυτά αποτελέσματα. Έχουμε δει κάποια πρόοδο να γίνεται. Πήγα στο Τσαπτσαράν στην ε, επαρχία Γκόρ και μου είπε και ένας αρχιεδικαστής ότι ένας ε, βαθμός και ένας εισαγγελέα ε, συνελήφθησαν ε, για λόγους διαφθοράς και επισκέφθηκα και τη μονάδα καταπολέμησης διαφθοράς στο Γενικό Εισαγγελέα όπου εργάζεται η UPOL και συνεργάζεται με τρεις εισαγγελείς και τους εκπαιδεύει τους Αφγανούς εισαγγελείς για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Υπάρχει λοιπόν μια προσπάθεια ε, και της διεθνούς κοινότητας ε, και για τη δικαιοσύνη και για την καταπολέμηση της διαφθοράς όσο γίνεται πιο εστιασμένα και βεβαίως με κριτήρια και προϋποθέσεις. Ε, ο αγαπητός φίλος Σελκύρης ρώτησε κάτι πολύ κρίσιμο αν θα κερδίσουμε, αν θα χάσουμε. Να σας πω κάτι, δεν μας παίρνει να χάσουμε. Είναι τόσα πολλά τα ζητήματα, είναι τόσο σκληρά τα ζητήματα, δεν ε, χωράνε εύκολες λύσεις, ούτε γρήγορες λύσεις. Ε, προχωράει ε, η πολιτική συμμετοχή και του χρόνου θα είναι ακόμα πιο έντονη και πιο ενισχυμένη. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα ότι είναι διαφορετική η χώρα, ότι έχουν δικές τους ε, ε, αξίες, δικές τους θρησκείες και θα πρέπει αυτό να τους σεβαστούμε. Αλλά όπως έδειξαν και οι προετοιμασίες για τις εκλογές, ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε με μια διαδικασία πιο συμμετοχικής δημοκρατίας και να σεβόμαστε και τις πραγματικότητες επιτόπου. Νομίζω ότι απάντησα για τις εκλογές, για τα διπλά κριτήρια ε, ναι, για το αφγανικό δίκτυο και τα διεθνή μέσα. Και το έχουμε καταγράψει αυτό. Αλλά τώρα η διαδικασία αυτή ε, είναι καθοδόν και ε, η Εφορευτική Επιτροπή θα πρέπει να απαντήσει ε, για τις καταγγελίες και τα παράπονα που έχουν κατατεθεί Και αυτό δεν είναι για μα, αλλά για να, πιστούν οι Αφγανοί οι ίδιοι ότι η διαδικασία είναι ε, διαφανής και σωστή. Γι' αυτό θα πρέπει και εσύ και το Μελλοντικό Κοινοβούλιο να αποκτήσουν ε, οντότητα θεσμών. Ο Πρόεδρος... Α, ο κύριος Σογόλτερ από τη Βρετανία έκανε μια ενδιαφέρουσα πρόταση με κάθε σεβασμό, εύκολα το λέτε, αλλά για να το κάνουμε και όλα αυτό στην πράξη. Ναι. Πήγαμε τον ε, δικό σας πρέσβη ε, με ελικόπτερο και πέταξα πάνω από τις καλλιέργειες και είδα τις καλλιέργειες της ε, ε Μύκονος, της Υπνοφόρου. Ωραία. τι να κάνουμε. μιλάμε για καινοτόμα προγράμματα, αλλά δεν είναι βιώσιμα, δεν είναι αηφόρα, δεν θα κάνουμε τίποτα. Έγιναν κάποιες απόπειρες, ε, αλλά δεν απέδωσε. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πολλά χρήματα για ε, εναλλακτικές καλλιέργειες για τη στήριξη εισοδήματος των αγροτών στη χώρα. Και νομίζω ότι απάντησα και κάτι διαφθορά σε αυτό. Και ένα τελευταίο, χωρίς αυτό είναι λιγότερο σημαντικό, ε, δικαιοσύνη. Βεβαίως, ε, είναι και πάλι πολλές οι του προβλήματος. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η διοικητική μηχανή είναι πάρα πολύ αδύναμη. Τους βοηθάμε. Είχαμε ένα εμπειρογνώμονα που βοήθησε να επανακαταρτιστεί το πρόγραμμα καλής χρηστής διακυβέρνησης όπως λέγεται ιδιαίτερα ως προς το δικαστικό σκέλος. Και τώρα έχουμε αναθέσει σε έναν άλλον εμπειρογνώμονα να μελετήσει τα θέματα με τρία δικαστικά, τρεις δικαστικούς θεσμούς. Ε, το, ε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, την Εισαγγελία και τους ε, δικαστές της έδρας, ας πούμε, τον αρχιδικαστή. Ε, και να τους δείξουμε τα βασικά, τις προτεραιότητες, τους βαθμούς, τις αμοιβέ, την ασφάλεια. Πώς να στηθεί ε, ε, μια δικαστική ε, εξουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Για έξι άτομα που έχουν ζητήσει το λόγο, παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Έχουν ήδη υποβληθεί πολλές ερωτήσεις και απαντήθηκαν. Ας αποφύγουμε τις επαναλήψεις. Πρέπει να τηρήσουμε απόλυτα το χρόνο μας. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη που είστε μαζί μας σήμερα εδώ το Αφγανιστάν είναι μια χώρα με συγκεκριμένες παραδόσεις που δεν έχουν ε, καμία, και καμία, κανένα παρελθόν κεντρικής κυβέρνησης, κεντρικής διακυβέρνησης. Πρόκειται να εγκρίνουμε ένα ψήφισμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλοί από εμά θέλουμε να εκφράσουμε τις πολιτικές απόψεις των λαών μας να φύγουμε από αυτή την παγίδα στην οποία έχουμε μπλακεί εδώ και 9 χρόνια και διερωτώ με ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την πρόταση να οργανωθεί μια πολιτική διαδικασία στο Αφγανιστάν η οποία θα συμπεριλάβει όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις με στόχο να μπορέσουμε να αποσύρουμε τις δυνάμεις του συνασπισμού μόλις αυτό καταστεί δυνατό. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό. Ποιος πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια τέτοια διαδικασία. Η άποψή μου είναι ότι πρέπει να φύγουμε από αυτή την παγίδα. Όσο περισσότερο μένουμε, τόσο πιο βαθιά θα βυθιστούμε μέσα σε αυτή την παγίδα. Και αυτό που δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο Αφγανιστάν είναι να γίνει ένας παράδεισος για την διεθνή τρομοκρατία όλα τα υπόλοιπα είναι ψευδέστηση. Δεν μπορούμε εμείς να διαχειριζόμαστε αυτή τη χώρα. Πρέπει εκείνη να αναλάβει τα ίνια τη διακυβέρνησή τη. Ο κύριο Ράιμα πρόεδρος Επιτροπής Άμυνας ε, του Κοινοβουλίου της Εστονίας. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου αφορά ένα θεσμικό όργανο, για ένα θεσμό, είναι το κοινοβούλιο, το, κοινοβούλιο του Αφγανιστάν, για το οποίο δεν ακούσαμε τίποτε. Υποστηρίζουμε την κεντρική κυβέρνηση και τις, επαρχε, και τις περιφερειακές κυβερνήσεις, την αστυνομία, το εκλογικό σύστημα στο Αφγανιστάν αλλά τι γίνεται με το κοινοβούλιο της χώρας αυτής. Πολλές φορές, έχω πάει πολλές φορές στο Αφγανιστάν και έχω επισκεφθεί και το κοινοβούλιο. Ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα υποστήριξης του Κοινοβουλίου του Αφγανιστάν από τεχνική άποψη στην Εθνία και καλώ τους συναδέλφους από τα άλλα κοινοβούλια να βρουν έναν τρόπο και αυτοί να υποστηρίξουν τους συναδέλφους βουλευτές του Κοινοβουλίου της, ε, του Αφγανιστάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω να ενισχύσουμε τη θέση του στα πλαίσια της κοινωνίας του Αφγανιστάν γιατί φοβάμαι ότι έχουμε την τάση να τους ξεχνάμε του βουλευτέ του Αφγανιστάν και αυτό είναι σημαντικό. Ο κύριος Τάνοκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο κύριο Ζήγκρι φαίνεται να, να διαρωτάτε ότι οι κοπέλες, οι κοπέλες εκπαιδεύονται στο Αφγανιστάν χωριστά από τα αγόρια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει, αυτό αποτελεί πρόβλημα. Το χειρότερο πρόβλημα είναι ότι σε ορισμένε περιοχέ τη χώρα δεν, έχουν, δεν λαμβάνουν την παραμικρή εκπαίδευση και ο ποινικό κώδικας περιλαμβάνει ορισμένες διατάξεις οι οποίες ευτυχώς δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής αλλά οι οποίες οπωσδήποτε προσβάλλουν τα δικαιώματα των γυναικών. Γίνονται αρκετές προσπάθειες για τον έλεγχο των ε, ε, υπηρεσιών πληροφορίας υποστηρίζοντας τους Ταλιμπάν και σε συνεργασία με τους Ταλιμπάν του Πακιστάν με κίνδυνο να αποσταθεροποιηθεί το Πακιστάν που προσπαθεί να συνέλθει από τις πλημμύρες και ποιος είναι ο ρόλος της ε, Ινδίας σε ό,τι αφορά τις ξένες άμεσες επενδύσεις και την ενίσχυση των θεσμών συνεργάζεται με την Ινδία και τέλος ποιες είναι οι εναλλακτικέ οδοί ε, φοδιασμού που θα παρακάμψουν το, το Πακιστάν ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια των δυνάμεων της ISAF και των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κιλ Νίλσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. το τελικό ανακοινωθέν της διάσκεψης της Καμπούλ προβλέπει ότι μέχρι το 2012 5% της παγκόσμιας ενίσχυσης θα περνάει μέσα από τον προπολογισμό του Αφγανιστάν. Μετά από την υπόθεση της Τράπεζας της Καμπούλ, τι προβλέπετε, τι σχεδιάζετε προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι αυτά τα κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν για σωστούς, για καλούς σκοπούς. Αυτή είναι το πρώτο μέρος της ερώτησή μου που συνδέεται και με όλα τα θέματα τη διαφθοράς που αναφέρθηκαν και θα ήθελα να έρθω και σε μια άλλη ερώτηση σχετικά με τη δουλειά των ε, δημοσιογράφων. Η πρόσβασή του σε ενημέρωση και σε πληροφορίε στη χώρα αυτή. Δύο δημοσιογράφοι Γάλλοι, ο Ερβέγγε Κέρ και ο Στεφάν Ταπονιέ, κρατούνται εδώ και εννέα μήνες στο Αφγανιστάν. Οι γαλλικές αρχές βεβαίως ανησυχούν για την τύχη τους και ενδιαφέρονται τακτικά για την κατάστασή τους, αλλά θα ήθελα αν είναι δυνατό, τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να ελευθερωθούν αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι. Merci. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φροντζουλίτσα από τη Ρουμανία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φαίνεται ότι είμαστε έγκλειστοι εδώ εξαιτία τη απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα βασικό θέμα, όπως την κατάσταση στο Αφγανιστάν. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον πρέσβη και να του ευχηθούμε κάθε επιτυχία στο έργο του. Βεβαίω είναι μεγάλη πρόκληση για τις χώρες μας. Αυτή η αποστολή δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Αλλά το Αφγανιστάν είναι μια ευκαιρία και για την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση έτσι ώστε να διαφημίσουμε μέσα σε εισαγωγικά και να βελτιώσουμε τις ικανότητές μας ως προς την ανοικοδόμηση και την διαχείριση κρίσεων. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε γιατί δεν υπάρχουν μόνο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες. Είναι και μία δοκιμασία ως προς τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ και ως προς τη βιωσιμότητα των διμερών σχέσεων. Ε, εφόσον το ΝΑΤΟ είναι πιο καλά εξοπλισμένο και διαθέτει διαφορετική πραγματογνωμοσύνη, εμείς θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην θεσμική ανάπτυξη. Έτσι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε στο Αφγανιστάν. Όταν μιλάμε για βιώσιμη συνεργασία, με όλους τους περιφερειακούς και διεθνείς εμπλεκόμενους φορείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, διότι η χρηστή διακυβέρνηση είναι ύψη τη σημασίας και θα πρέπει να την προωθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αφγανιστάν, διότι πέρα από το να νιώθει κανείς ασφαλής, οι κάτοικοι του Αφγανιστάν θα πρέπει να ξέρουν ότι μπορούν να ε, βασιστούν σε θεσμικά όργανα τα οποία ε, επικεντρώνονται στους πολίτες και στα συμφέροντα των ε, πολιτών. Μετά από αυτά τα σχόλια, τα προκαταρκτικά, θα ήθελα να, πω πώς βλέπετε, να ρωτήσω πώς βλέπετε την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών, διότι το 2011, το δεύτερο εξάμεινο του 2011, ορισμένες χώρες ανακοίνωσαν ότι θα αποσύρουν τα στρατεύματά τους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάννης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξοχότατε κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σας και για την παρουσίασή σας. Ο κύριος Χαβιέρ Σολάνα, την περασμένη Παρασκευή, προχθές δηλαδή, ε, στην παρουσίαση ενός βιβλίου που μόλις δημοσίευσε, είπε στη Μαδρίτη ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν ήταν αδύνατο να κερδιθεί στρατιωτικά. Γιατί ξέρουμε και από πού προέρχεται ο κύριος Σολάνα και τη δήλωση είναι αυτή. Εσείς τι λέτε γι' αυτό. Και επειδή ο φίλος ε, Νταντζάν έχει προβλήματα με το χρόνο, δεν θα πω άλλα. Ε, απλώς να έχετε υπόψη σας ότι είμαι από εκείνου που πιστεύουν ότι σχεδόν τα πάντα είναι καλύτερα από να επιτρέψει η ε, διεθνής κοινότητα να έρθουν στην εξουσία οι Ταλιμπάν και να ε, καταδυναστεύουν το λαό και να ξαναγίνει το Αφγανιστάν ένα νέο ε, άνδρο και άσυλο για τη διεθνή τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Ξεχώτατε. 10 λεπτά παρακαλώ. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες και προκλητικές ερωτήσεις. Κύριε Τάλερ, για να απαντήσω στον ε, κύριο Τάλερ καταρχήν και σε σχέση με την ε, πολιτική διαδικασία. Η απάντηση, δεν μπορεί, η απάντηση είναι ότι ο πόλεμος, μάλλον μας είπατε, ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί στρατιωτικά. Μα βρισκόμαστε σε μία ε, διαδικασία εξελικτική Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της αφγανικής κυβέρνησης για τη συμφιλίωση. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε, όπως είπε και ο κύριος Τάλερ, ότι η απόσυρση είναι δυνατή μόνο όταν δημιουργήσουμε τα θεμέλια έτσι ώστε οι Αφγανοί να μπορέσουν να διακυβερνήσουν τη χώρα τους. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο γι' αυτό, επαναλαμβάνω, όπου συναντώμε με το κοινό και με τα ΜΜΕ. Αν φύγουμε τώρα θα αφήσουμε μία αναστάτωση πίσω μας, θα ενισχυθεί η τρομοκρατία και θα οδηγήσει σε περιφερειακή αστάθεια αν όχι σε πόλεμο. Γι' αυτό θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλους όσους συνεισέφεραν για την πολιτική σταθερότητα στο Αφγανιστάν και ιδιαίτερα για τους πεσόντες πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε μόνο στρατιωτικά, θα πρέπει να προβάλλουμε και πολιτικές ικανότητες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Σε σχέση με το ερώτημα του ε, Εσθονού Προέδρου της Επιτροπής, Εθνικής Επιτροπής Άμυνας, ε, υποστηρίζω αυτό που είπατε, δηλαδή τα προγράμματα υπέρ της κυβέρνησης του Αφγανιστάν. Αυτό το έχω συζητήσει και με το προσωπικό της, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτό το εφαλτήριο, αυτή την όθηση και επειδή Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου θα συγκροτηθεί νέα κυβέρνηση. Θα πρέπει να τους καθοδηγήσουμε για να γνωρίσουν πώς λειτουργεί ένα κοινοβούλιο, ποιες είναι οι σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Γι' αυτό έκρινα ότι θα πρέπει να μεταβούμε, να επισκεφθούμε το νέο κοινοβούλιο του Αφγανιστάν και να προωθήσουμε τις διακοινοβουλευτικές σχέσεις όπως ζήτησα από τον πρόεδρο Μπούζεκ. Σε σχέση με την εκπαίδευση, με αυτό το σκέλος δεν θα ήθελα να το σχολιάσω τόσο πολύ ο Βρετανός βουλευτής ε, μίλησε για το Πακιστάν. Ο κύριος Τάνοκ αναφέρθηκε σε αυτό. Καταλαβαίνουμε την συνδεσιμότητα, την, μάλλον ε, αυτή την, τη σύνδεση αυτών των δύο χωρών και ξέρουμε πως έχει και η τρέχουσα κατάσταση. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί προγράμματα και στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν και εγώ έχω μεταβεί στο Ισλαμαμπάτ καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς τα Ηνωμένα Έθνη και είδαμε να επιτελείται πρόοδος της διμερής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών. Χρειάζεται επικοδομητική συνεργασία για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την διασυνοριακή τρομοκρατία. Ιδιαίτερα ως προς το Αφγανιστάν-Πακιστάν. Σε σχέση με τις εναλλακτικέ οδούς, με τα εναλλακτικά μέσα, υπάρχει έλεγχος στις παραμεθόριους περιοχές Πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν εναλλακτικέ για τον, ε, για τον έλεγχο μεταξύ Αφγανιστάν, Πακιστάν και Κεντρικής Ασίας. Επίσης είδαμε ορισμένα ενθαρρυντικά σημάδια συνεργασίας στα πλαίσια της ευρύτερης ε, περιοχής, ιδιαίτερα ως προς τον αγωγό φυσικού αερίου που περνάει από το Τουρκμενιστάν και φτάνει στην Ινδία. Έτσι, θα δημιουργηθεί μια νέα πλατφόρμα οικονομικής συνεργασίας και διασύνδεσης μεταξύ αυτών των χωρών, διότι και οι Πακιστανοί έχουν επενδύσει πολύ στο Αφγανιστάν. Έτσι ώστε να μην υπάρχουν αντιπαλότητες και ρήξεις. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί μπορεί να προσπαθεί να διαμορφώσει αυτή τη διεθνή ατζέντα μέσα στα πλαίσια της ΡΕΚΑ, της Περιφερειακής Διάσκεψης Συνεργασίας στο Αφγανιστάν. Στις 3 και 4 Νοεμβρίου θα συνεδριάσει η ΡΕΚΑ για να, όπου θα γίνει λόγος σε αυτή τη διάσκεψη για τους διασυνοριακούς ελέγχους. Το συζήτησα με τους πρέσβεις του Πακιστάν και της Ινδίας. Και με τον τελευταίο παίζουμε και τένις. Τώρα, πώς μπορούμε να προωθήσουμε περαιτέρω ε, χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της ε, κατάστασης και τη διοχέτευση χρημάτων στην Καμπούλ. Εγώ ήμουνα επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με τις αφγανικές αρχές. Βεβαίως θα ε, χορηγήσουμε αυτές τις, ε, αυτή την ενίσχυση μόνο όμως αν καταπολεμηθεί η διαφθορά. Αυτό το είπαμε και στο, προς τον πρόεδρο Καρζάη και στις αφγανικές αρχές. Δεν θα ήθελα να πω σε λεπτομέρειες ως προς τα θέματα των δύο δημοσιογράφων. Είναι, βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων μεταξύ αφγανικών και γαλλικών αρχών. Ο Ρουμάνος βουλευτής υπέβαλε ένα ερώτημα για το τι θα γίνει στο τέλος του 2011 όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις ε, θα αποδυναμωθούν, θα μειωθούν. Αναφέρεστε στη Γιούπολ, αν καταλαβαίνω καλά, γιατί όλα, τα υπόλοιπα θέματα αφορούν τον ΝΑΤΟ και ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος ε, ε, Ράσμουσεν, θα επεκταθεί επί αυτού του θέματος. Ως προς την πολιτική αστυνομία ελπίζουμε να μπορέσει να συμμετάσχει πιο ενεργά σε αυτή την μεταβατική περίοδο και να δράσει ακόμα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους. Ο Γενικός Γραμματέας ΝΑΤΟ κύριος Ράσμονσον θα είναι εδώ σε λίγα λεπτά. Διακόπτουμε και θα ξαναρχίσει η συνεδρίασή μας στις 4. Θα ήθελα να επαναλάβω ακόμα μια φορά σε όλους τις ευχαριστίες μου για τον ενδιαφέρον που δείξατε στο Αφγανιστάν. Αυτό θα με βοηθήσει στις μελλοντικές ε, δραστηριότητες μου στην Καμπούλ για την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ βρίσκεται μεταξύ μας στην ώρα του και θα θέλαμε και εμείς να ανταποκριθούμε αρχίζοντας τις εργασίες μας εγκαίρως. Θα ήθελα εξ ονόματος όλων να σας ευχαριστήσω γιατί δεχτήκατε να συμμετέχετε στις εργασίες μας και να μας ενημερώσετε ως προς την κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Μιλάμε για μία νέα και πολύ σημαντική εξέλιξη. Πέρα από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της ε, Λισαβόνας και το αποτέλεσμα αποτύπωμα που άφησε στην ΕΠΑ υπάρχει και γίνεται μάλλον μια σημαντική συζήτηση σε επίπεδο ΝΑΤΟ για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές και την γενικότερη στρατηγική και προτεραιότητες ως προς τις παρεμβάσεις για τα μελλοντικά έτη. Πέραν από τους εκπροσώπους ευρωβουλευτές έχουμε και εκπροσώπους από τα Εθνικά Κοινοβούλια και ιδιαίτερα από τις Επιτροπές Άμυνας και Ασφάλειας ή Επιτροπές Ευρωπαϊκών Σχέσεων. Υπάρχουν ε, θέματα που άπτονται των εργασιών και αυτών των επιτροπών και αφορούν όλους τους πολίτες. Όπως ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινούς στόχους με το ΝΑΤΟ, δηλαδή να προωθήσουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα στις, ε, στην περιφέρειά μας, αλλά και πέραν αυτής. Γι' αυτό ξέρετε, όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, 21 από τα 27 κράτη-μέλη είναι μέλη και του ΝΑΤΟ. Και γι' αυτό συνεργαζόμαστε ως προς τους ε, στρατιωτικούς στόχους και την στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ. Μπορούμε να αναφερθούμε στο Κωσυφοπέδιο και το Αφγανιστάν για τις κοινέ μας επιχειρήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και την θέση σε ισχύ Τη συνθήκη της Λισαβόνας με μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Θα πρέπει λοιπόν να εξεύρουμε διαφορετικές και πιο αποτελεσματικές μεθόδους συνεργασίας και συμμιλωματικότητας ως προς τις ε, σχέσεις μας και τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Είχα αναφερθεί στην αρχή στο γεγονός ότι το ΝΑΤΟ ε, διανύει μια φάση περί συλλογής ως προς τη λειτουργία και το επιχειρησιακό του πλαίσιο. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε ποιες είναι οι κατευθυντήριες γραμμές που θα προτείνετε στα μέλη της Συμμαχίας στις 14 Οκτωβρίου, διότι προβλέπεται συνάντηση με τους Υπουργούς Εξωτερικών επί του θέματος αυτού. τον ε, Ιούλιο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μαζί σας και πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την διαδικασία ε, μεταρρύθμισης ε, μέσα στα πλαίσια μιας αγαστής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας δίνω το λόγο κύριε Γενική Γραμματέα. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη θερμή σας υποδοχή και την ευγενή σας εισαγωγή. Είμαι ε, πολύ ευτυχής ε, που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι και πάλι ενώπιον σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ε, απευθύνομαι ταυτόχρονα σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και σε μέλη εθνικών κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλησα να έρθω στο κοινοβούλιο σας για να ανταλλάξουμε απόψεις και να σας ζητήσω να υποστηρίξετε την φιλοδοξία μου να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ με τρόπο ουσιαστικό. Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση γνώρισαν βαθύτατες αλλαγές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ πρόσφατα άλλωστε με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταγωνιστή σε πολλά επίπεδα εγνωσμένου κύρους ε, στη διεθνή σκηνή, συμπεριλαμβανομένων και των θεμάτων αμήνης, γιατί ηγείται σε πολλές ε, πολιτικές αποστολές και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε διάφορες ε, κονίστρες στο εξωτερικό της. Μια συνεργασία λοιπόν στενότερη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ε, κατέστη πλέον στρατηγική ανάγκη. Θα ήθελα καταρχάς να πω δύο λόγια ως προς την οργάνωση, τον οργανισμό μάλλον που έχω το προνόμιο να ηγούμε. Το σημερινό ΝΑΤΟ είναι πολύ διαφορετικό από τη συμμαχία ε, του ψυχρού πολέμου. Βεβαίω, οι θεμελιώδεις αρχές δεν έχουν αλλάξει. Διατλαντική συμμαχία με στεναρή προσήλωση στην αμοιβαία ε, υπεράσπιση άμυνα απέναντι σε κάθε απειλή και κάθε επίθεση και όπου όλα τα κράτη-μέλη του οργανισμού ε, προσιλώνονται και στενίζονται τις ιδέες που μας είναι τόσο προσφυλείς. Νέο στρατηγικό δόγμα. Θα ε, καταρτιστεί στη Λισαβόνα το Νοέμβριο, στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ. Και αυτό θα είναι σημαντική φάση, σημαντικό στάδιο ε, στην προσαρμογή της συμμαχία. Αυτό το νέο λοιπόν στρατηγικό δόγμα θα είναι το όραμά μα, αλλά και ο καθοδηγητής μας για την επόμενη δεκαετία και θα ορίσει και το δρόμο που θα ακολουθήσουμε για να δώσουμε νέα δυναμική και να ενισχύσουμε τη συμμαχία. Θα είναι λοιπόν μια στρατηγική για το ΝΑΤΟ ταυτόχρονα εφικτή αλλά και βιώσιμη. Υπό την έννοια αυτή, χθες υπέβαλα ένα σχέδιο κειμένου στους συμμάχους, μέλη ε, του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Οι σύμμαχοι θα διαπραγματευθούν ε, το τελικό κείμενο κατά τη διάρκεια των ερχομένων εβδομάδων. Το στρατηγικό μας δόγμα θα βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες. Πρώτον, στα αγγλικά τώρα. Ασφάλεια και άμυνα στον 21ο αιώνα. Η προσήλωσή μας για συλλογική άμυνα βάσει του άρθρου 5 είναι στεναρότατη και θα την υποστηρίξουμε με τις ανάλογες στρατιωτικές δράσεις. Επίσης θα ε, ασχοληθούμε με το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε νέες ε, ε, προκλήσεις και απειλές, όπως είναι απειλές στον κυβερνοχώρο, με διάδοση μέσω μαζικής καταστροφής, τρομοκρατία και διατάραξη διακοπή του ανεφοδιασμού μας σε ενέργεια. Δεύτερο, ασφάλεια μέσω διαχείρισης των κρίσεων αντί να αντιδρούμε σε συνέπειες των κρίσεων, αυτή τη στιγμή έχει ξεσπάσει η βία, θα πρέπει να είμαστε προληπτικοί, συγγνώμη, να δρούμε προληπτικά ε, σε πρώιμα στάδια για να συντονίζουμε καλύτερα τις δράσεις μας με άλλους οργανισμούς που επιφορτίζονται με τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό ε, το ονομάζουμε συνολική προσέγγιση. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε τις σωστές ικανότητες αλλά και σχέσεις για να το κάνουμε αυτό. Τρίτον, πώς μπορεί να προωθήσει το ΝΑΤΟ τη διεθνή σταθερότητα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη συνέχεια θα επεκταθώ στις προτάσεις ε, που κάνω για το σκοπό αυτό. Ήταν πραγματική επιτυχία ε, οι πολιτικές του ΝΑΤΟ για συνεργασία με ε, χώρες και με άλλους οργανισμούς και θα πρέπει να επενδύσουμε εκεί με περισσότερο διάλογο, περισσότερη συνεργασία με χώρες ανά τον κόσμο, χώρες οι οποίες ε, μοιράζονται το δικό μας συμφέρον στο να υπάρχουν ειρηνικές διεθνείς σχέσεις συμπεριλαμβανομένων κρατών όπως είναι η Ινδία και η Κίνα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να διευρύνουμε το φάσμα των θεμάτων που είμαστε διατεθειμένοι να συζητούμε με τις χώρες αυτές με τις οποίες διατηρούμε σχέσεις, καθώς και με άλλους οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη. Τέταρτον και τελευταίο στοιχείο στο νέο στρατηγικό μας δόγμα είναι ο μετασχηματισμός και η μεταρρύθμιση του ΝΑΤΟ. Η μεταρρύθμιση είναι μια διαδικασία διαρκής και όχι στιγμιαία. Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικά καιρούς το στρατηγικό δόγμα θα πρέπει να ανοίξει ένα δρόμο έτσι ώστε να αποδίδει περισσότερο ε, ο αμυντικός προπολογισμό και να μας ε, εξασφαλίζει και περισσότερη προστασία, καλύτερη ασφάλεια. Τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να αναπτύξουμε καλύτερα τις δυνάμεις μας, αλλά παραμένουν ε, σε στρατόπεδα που είναι απόρρια του ψυχρού πολέμου ε, ακριβά στη συντήρησή του και δεν ξέρουμε τι ακριβώς να τα κάνουμε. Για ποιο λόγο θα διατηρούμε αυτά ακόμα. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Επιτρέψτε μου να εστιάσω σε ένα ιδιαίτερο θέμα που θα κυριαρχήσει στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας. Εν ώψη της απειλής που συνιστά η διάδοση των πυράβλων, θα πρέπει καλύτερα να προστατευθούμε. Η Συμφωνία για Ανάπτυξη μια δυνατότητας ε, αντιπυραυλική προστασίας ε, υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ θα μας βοηθήσει να το κάνουμε αυτό και αν υπάρξει συμφωνία να επεκταθεί το σημερινό πρόγραμμα, το οποίο σήμερα προστατεύει μόνο τις ε, ένοπλες δυνάμεις μας σε ανάπτυξη. Λοιπόν, εφόσον επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσαμε να δίνουμε αντιπυραυλική κάλυψη και ε, στην επικράτεια και στους λαούς των Ευρωπαίων μας συμμάχων. Δηλαδή, να ε, συνδεθεί όχι μόνο με την ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών μας, αλλά και με συγκεκριμένη επικράτεια αυτό το αντιπυραυλικό μας σύστημα. Επανέρχομαι στη συνολική αυτή προσέγγιση σημερινή, οι σημερινές απειλές και οι προκλήσεις είναι πολύπλευρες, είναι πολυμερείς και ιδιαίτερες και περίπλοκες και χρειάζεται πολιτική συνεργασία, στρατιωτική, οικονομική και άλλα μέτρα αλληλοσυμπληρούμενα. Το ΝΑΤΟ έχει την ισχύ του και ε, ε, τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι παράγοντες και φορείς όπως είναι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Για να βεβαιωθούμε λοιπόν ότι αυτές οι δυνάμεις αλληλοενισχύονται θα πρέπει να συνομιλούμε, να διδασκόμεθα ένας από τον άλλον και να δρούμε και από κοινού όταν αυτό έχει νόημα. Στη δεκαετία του 90, όταν συνενώθηκε η ε, διατλαντική κοινότητα για να τερματίσει τη σύραξη στα Βαλκάνια, είχαμε ε, ελπίδες ότι θα διευρυνθεί αυτή η συνεργασία. Ενώ έγινε μια καλή αρχή, δυστυχώ δεν καταφέραμε να οικοδομήσουμε ε, πάνω σε αυτό και να αναπτύξουμε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων ασφαλείας που να διαπραγματευόμαστε. Για ποιο λόγο, για να το πω απλά. Οι εθνικές αντιλήψεις για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ διαφέρουν και εξακολουθούν να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Ορισμένες χώρες θέλουν να υπάρχει στενή σχέση ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και αυτό το ε, θέτουν ως πολιτική προτεραιότητα. Άλλες διστάζουν και παραμένουν διστακτικές και ε, δηλώνουν ότι η στενότερη σχέση μπορεί να υπονομεύσει τη σχέση των δύο οργανισμών ή μπορεί να εισαγάγει κάποιο είδους ιεραρχία στις σχέση τους. Θέλω να καθησυχάσω εκείνους που διστάζουν ότι το ΝΑΤΟ σέβεται την αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λήψη των αποφάσεων. Βεβαίω και διατηρεί και τη δική του αυτονομία στη δική του λήψη αποφάσεων. Επιπλέον, ευρύτερη συμμαχία στρατηγικής φύσεως σημαίνει ότι και οι δύο εταίροι συνεργάζονται επίσης όρει. Πράγμα προαπαιτούμενο για μια ε, σχέση αμοιβαία εμπιστοσύνης τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει πολλές προτάσεις μέλη και των δύο οργανισμών για να μας φέρουν πιο κοντά. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία ε, και να επιταχύνουμε και να αναβαθμίσουμε τη συνεργασία μας στους εξής τρεις βασικούς τομείς. Πρώτο και σημαντικότερο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ χρειάζεται να έχουν τακτές, τακτικές επαφές ε, σε όλα τα επίπεδα, σε όλο το φάσμα των κοινών ενδιαφερόντων μας για την ασφάλεια. Σήμερα ε, ζούμε μια ατυχή κατάσταση. Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να συζητούν επισήμω σημαντικά ζητήματα, αλλά πλην της Βοσνίας. Παρά το γεγονός ότι μοιραζόμαστε πολλά ε, ε, συμφέροντα ασφαλεία σε πολλού τομεί. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνεργάζονται πιο στενά στις επιχειρήσεις. Όλο και περισσότερο συναντάμε ένα τον άλλον ε, σε διεθνείς καταστάσεις στο στη, στο Αφγανιστά και στα ανοιχτά των ακτών της Σομαλίας. Και οι δύο οργανισμοί έχουν διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή του, αλλά θα πρέπει να είναι συμπληρωματική η προσέγγιση. Για να γίνει αυτό χρειάζεται συντονισμό άλλου επίπεδου. Και ένα τρίτο, ο αμυντικό προπολογισμό θα πρέπει να πιάνει περισσότερο τόπο. Παράδειγμα, ένα και μόνο. Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε μια κοινή προσέγγιση αναπτύξει για να αντιμετωπίσουμε τους λεγόμενους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς και μάλιστα οργανισμούς που βάζουν στην άκρη των δρόμων και αυτό κοστίζει πολλές ε, ζωές πολιτών και στρατιωτών στο Αφγανιστάν. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορούμε από κοινού να αποφύγουμε επικαλύψεις και να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους που είναι και ε, περιορισμένοι πιο αποτελεσματικά. Για να ξεπεράσουμε λοιπόν τις πολιτικές δυσκολίες, ε, πρότεινα μια διτή προσέγγιση όταν συνήντησα τους Υπουργούς Αμήνης στην Πάλμα Μαγιόρκα τον περασμένο Φεβρουάριο αμήν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η μία πλευρά. Και από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τους συμμάχους που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα πολιτικά και στρατιωτικά. Και συγκεκριμένα έθεσα τα εξής τρία ζητήματα. Πρώτον, καλύτερη συμμετοχή συμμάχων που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα και δραστηριότητες κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει στην Τουρκία μια συνολική συμφωνία ασφαλείας Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμφωνήσει ε, να ε, υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης. Αυτά τα επέβαλα και υπόψη του Προέδρου Μπούζεκ και σε πολλούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, χάρηκα από τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πριν από δύο εβδομάδες και προσβλέπω συνεργασία με την κυρία Άστον για να λύσουμε τις πολιτικές διαφορές που είναι εμπόδιο ενδεχομένω ε, στη συνεργασία ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε δέσμευση στα ε, υψηλότερα κλιμάκια τη πολιτική για να προχωρήσουμε. Ιδιαίτερα οι 21 χώρε που είναι μέλη και των δύο οργανισμών μπορούν και οφείλουν, πιστεύω, να διαδραματίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ε, αναζήτηση λύσεων. Συμπερασματικά, γνωρίζω πάρα πολύ το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχω επίγνωση και Γι' αυτό προσβλέπω στην υποστήριξή σα και περιμένω να ακούσω και τι αντιδράσει σας στις ε, πολλές προτάσεις που έκανα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Γενική Γραμματέα. Η παρέμβασή σας ήταν πλήρης, κέρια και στα χρονικά περιθώρια τα οποία ας πούμε είναι αποδεκτά για να μπορέσουμε να προωθήσουμε μία συζήτηση αρκετά διεξοδική. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Ντανζόν, στον πρόεδρο της Υποεπιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, ευχαριστούμε για το μήνυμά σας και για την παρουσία σας και απόψε εδώ. Ξέρετε ότι αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το διάλογο με τον ΝΑΤΟ. Η παρουσία σας, η τακτική παρουσία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Έχω δύο ερωτήσεις, πολύ σύντομε και ίσως όχι πολύ ευχάριστες. Η πρώτη που θα ήθελα να θέσω αφορά τις περίφημες πολιτικές ικανότητες στην σφαιρική προσέγγιση, comprehensive approach που θέλει να αποκτήσει το ΝΑΤΟ. Θεωρώ ότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις μεταρρύθμισεις, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προϋπολογισμού, γραφειοκρατίας, προσωπικού που θέλει να πραγματοποιήσει παράλληλα το ΝΑΤΟ. Πώς θα πετύχετε, θα ανταποκρίνετε σε αυτή την πρόκληση, πώς θα πετύχετε αυτό το στόχο να διευρύνετε τις ικανότητες σε πολιτικό επίπεδο του ΝΑΤΟ, ενώ περιορίζετε μέσα από μια ουσιαστική μεταρρύθμιση τα, για να αντιμετωπίσετε τα δημοσιονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός. Δεύτερο θέμα η Τουρκία. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο διάλογος, ο πολιτικός και σε θέματα ασφάλειας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ είναι σημαντικός. Αναφερθήκατε σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο Πέδιο, στο Αφγανιστάν και είπατε ότι ο μόνος διάλογος που μπορεί να έχουμε με την Βοσνία δεν αρκεί δέχομαι τις παραχωρήσεις που μπορούν να γίνουν στην Τουρκία και το διάλογο που μπορούμε να έχουμε σε θέματα ΕΠΑ με την Τουρκία, ωστόσο διαρωτώ με κατά πόσο παραχωρήσεις μόνο στην Τουρκία θα συμβάλλουν στη βελτίωση του διαλάγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Πρέπει να ισχύσουν ορισμένες ε, προϋποθέσεις έναντι των συναδέλφων της Τουρκίας. Η εξωτερική πολιτική έρχεται όλο και περισσότερο σε αντίθεση με δεσμεύσεις, παραβιάζει δεσμεύσεις που είναι οι ελάχιστες δεσμεύσεις ε, αλληλεγγύη στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Βεβαίως ένας διάλογος με την Τουρκία, ένας ενισχυμένος διάλογος με την Τουρκία και σε θέματα ασφάλειας, αλλά ένας διάλογος που θα είναι ταυτόχρονα και απαιτητικό. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο Ντανζόν. Πριν ε, ξεκινήσει η συζήτηση, θα ήθελα να καλωσορίσω μία ομάδα φοιτητών, είναι περίπου 70, που αποφύτησαν από, το, από την Ευρωπαϊκή Σχολή Άμυνας και Ασφάλειας και είναι εδώ παρόντες. Υπάρχει πληθώρα παρεμβάσεων. Θα ήθελα να αρκεστείτε στα τρία λεπτά έτσι ώστε να μπορέσετε να παρέμβετε όλοι και να απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας. Ο κύριος Τσουρκάσχη έχει το λόγο από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Βουλγαρίας. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα. Σας ευχαριστώ που ε, παρευρίσκεστε εδώ και μπορούμε να προωθήσουμε μια ουσιαστική συζήτηση Μέχρι τώρα είχαμε τη δυνατότητα να σχολιάσουμε την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι ένα δύσκολο ζήτημα και όπως μας είπε ο ειδικό εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν, οι προσπάθειές μας εστιάζονται στην ενίσχυση του πολιτικού σχεδιασμού, δηλαδή στην εκπόνηση ενός σωστού ε, διοικητικού συστήματος στο δημόσιο τομέα. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι αυτό που έχει σημασία είναι η κατάρτιση των αστυνομικών δυνάμεων και των στρατιωτικών για να μπορέσουν να αναλάβουν την διαχείριση των επιχειρήσεων επιτόπου. Πώς διαβλέπετε αυτή τη δυνατότητα δηλαδή να συντονιστούν οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του και του ΝΑΤΟ έτσι ώστε να έχουμε συμπληρωματικό χαρακτήρα και να μπορέσουμε να θέσουμε τέλος σε αυτή την σύραξη στο Αφγανιστάν. Μιλήσαμε και για το Πακιστάν. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι και η συμμετοχή της Ρωσίας. Ο Μετβέτεφ ε, διοργάνωσε ένα φόρουμ λίγους μήνες πριν και ο προκάτοχός σας, ο Λόρδος Ρόμπερτσον, παρευρέθηκε σε αυτό το φόρουμ για συζητήσεις. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η απαρχή μιας συμφωνίας μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας για να υποστηρίξει η Ρωσία συγκεκριμένους διαδρόμους διέλευσης. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα αποφασιστικότητα σε σχέση με, τη, με μια λήψη απόφαση σε, αυτό το, αυτή τη σύραξη αποφασιστικού χαρακτήρα στο Αφγανιστάν. Ο κύριος Λίζεκ έχει το λόγο. Ε, αντιπρόεδρος της Υποεπιτροπής Άμυνα και Ασφάλειας για τρία λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, το ΝΑΤΟ είναι ο θεματοφύλακας της ασφάλειάς μας. Αυτό αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές χώρες του κόσμου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, κάτι κύριε Γενικέ σε σχέση με τις χώρες που δεν νιώθουν ασφαλείς διότι δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Αν και οι χώρες αυτές είχαν εκφράσει την επιθυμία συμμετοχής. Δηλαδή μιλώ για την Γεωργία και την Ουκρανία. Η κατάσταση είναι πολύ δυσχερής σε αυτές τις δύο χώρες, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς δεχτήκατε την απόφαση του Προέδρου της Ουκρανίας που αναβάλει αυτή την πιθανότητα προσχώρησης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Όπως ε, ξέρουμε η κατάσταση δεν είναι καθόλου ε, απλή. Υπάρχουν ε, αντιμαχόμενες δυνάμεις. Υπάρχει και το κίνημα της Γιούλια Τιμοσέγκο, της πρώην Πρωθυπουργού, η οποία θέλει να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη προσχώρηση στο ΝΑΤΟ. Στη Γεωργία η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη μετά την ε, σύραξη το 2008. Όμως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το ότι οι πολιτικές δυνάμεις, κυβέρνηση και αντιπολίτευση όλοι είναι ομόφωνοι ως προς το ότι η Γεωργία θα έπρεπε να συμμετάσχει στις ε, δομές και δραστηριότητες του ΝΑΤΟ. Πώς ε, διαβλέπετε αυτή την κατάσταση, πώς αποτιμάτε αυτές τις πρόπτικες της Γεωργίας ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε. Έχουμε και ορισμένους άλλους ε, συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο και θα πρέπει δυστυχώς να περιορίσω το χρόνο σε δύο λεπτά για τους επόμενους ομιλητές. Δυστυχώς πρέπει να το επιβάλλω αυτό έτσι ώστε να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Ο κύριος Τζιγκάρης, προ... ε, συγγνώμη, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων από τη Λιθουανία. Έχετε λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Γενική Γραμματέα, είμαστε πολύ ευτυχείς που επιτέλους στείλατε ένα σημαντικό έγγραφο χθε στις εθνικές κυβερνήσεις και στα εθνικά μας κοινοβούλια, ώστε να εγκρίνουμε μια κοινή στρατηγική μαζί σας. Αλλά τα νέα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουν την παρουσία του ΝΑΤΟ στο χώρο τους. Βεβαίως, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που αναφερθήκατε στην πέμπτη παράγραφο και στην πρώτη υποχρέωση του ΝΑΤΟ, αλλά υπάρχουν άλλα σχέδια για το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε μαζί διότι προσχωρήσαμε πρόσφατα στο ΝΑΤΟ και χρειαζόμαστε μια πιο, πιο σαφή παρουσία για να προχωρήσουμε. Τι μέτρα λοιπόν κατά την άποψή σας θα έπρεπε να ληφθούν ώστε η παρουσία του ΝΑΤΟ να καταστεί πιο ορατή στις χώρες μας, στην περιοχή της Βαλτικής ειδικότερα όπου υπάρχει μόνο μία μονάδα αεροσκαφών και πώς θα μπορούσαμε να την ενισχύσουμε ώστε να αποκτήσει και μία μονιμότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοπά έχει το λόγο για δύο λεπτά. Thank ε, Σας ευχαριστώ. Κύριε Ράσμονσεν, θα ήθελα να μιλήσω μετά από τους συναδέλφους για την ιδέα του ΝΑΤΟ να προχωρήσει προς την ανάπτυξη δικών του ικανοτήτων στον τομέα της διαχείρισης κρίσεων. Για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτή θα είναι μια διπλοποίηση, επικάλυψη προσπαθειών εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός παίκτη σε αυτό τον τομέα. Σε τι βαθμό πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία τελικά θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σύμπραξη ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτικοστατιωτική συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θα μπορούσαν να προσφέρουν τις πολιτικές ικανότητες όταν οι δύο οργανισμοί επιχειρούν στην ίδια περιοχή κρίσεων. Θα ήθελα να επαναλάβω από την άποψη αυτή ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο υποστηρίζει την θέση ότι οποιαδήποτε ρήτρα συνεργασίας δεν πρέπει να γίνει σε βάρος της ανεξάρτητης ανάπτυξης των ικανοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να σέβεται τις υποχρεώσεις ουδετερότητας ορισμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κόπα. Ο κύριος Νεοφίτου, παρακαλώ, πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και εσείς έχετε τονίσει, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει ε, συμφωνήσει πως χρειάζεται να ενταθούν οι προσπάθειες για ενίσχυση της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα και μετά την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνα. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα ε, στις σχέσεις ε, ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια ειδική επιτροπή υπό την πρώην Υπουργό Εξωτερικών της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών, της κυρίας Ολπράιτ, είχε κάνει μια ανάλυση και εισηγήσει από το κρουπ των εμπειρογνωμόνων για ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο για τον άτομο και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην εισήγηση ότι full complementarity between NATO and the European Union will be essential. It should be noted, however, that full complementarity is only possible. Όμως ο συμπληρωματικός χαρακτήρας είναι δυνατός τη στιγμή που τα κράτη-μέλη που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ και αυτά που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ ε, έχουν έχουν πρόσβαση στις κοινέ δραστηριότητες. Του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ σε αυτή την εισήγηση υπό την Επιτροπή της κυρίας Όλπραϊτ. Η κυρία Γιαννάκου έχει το λόγο για δύο λεπτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ για τη σημερινή του παρουσία ε, οι ερωτήσεις είναι δύο πολύ σύντομες. Η πρώτη είναι ποιες είναι κατά το Γενικό Γραμματέα οι πραγματικές απειλές για την ασφάλεια των μελών του ΝΑΤΟ. Οι πραγματικές απειλές της σήμερα. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά στο Αφγανιστάν. Βλέπουμε ότι το Αφγανιστάν από πλευράς λειτουργίας δημοκρατικών θεσμών ε, έχει μια πολύ αρνητική κατάσταση ελπίζει ο Γενικός Γραμματέα ότι θα φύγει ποτέ από τον το ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν και θα είναι σε θέση το σύστημα να διατηρήσει μόνο τη δημοκρατία ή η προσπάθεια δεν θα έχει αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αρλάκη που είναι η συγητής για το Αφγανιστάν από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κύριε Γενικέ Γραμματέ, ευχαριστώ πολύ. Είναι η δεύτερη φορά που σας ακούω σε αυτή την Επιτροπή και πρέπει να πω ότι θαυμάζω την επιμονή και το πάθος σας όταν αμήνεστε υπέρ του ΝΑΤΟ και προσπαθείτε να μας πείσετε ότι έχει ακόμα πολύ σημασία και ότι αξίζει ακόμα να υπάρχει το ΝΑΤΟ και ορισμένες φορές μας πείθεται, αλλά άλλες όχι. Παραδείγματος χάρη, πρώτη ερώτηση. η εγκληματικότητα, η τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο. Σημαντική απειλή για την οποία χρειαζόμαστε τον ΝΑΤΟ για να μα υπερασπιστεί. Προσπαθήστε να με πείσετε πρώτον ότι οι επιθέσει στον κυβερνοχώρο είναι πραγματικά τόσο επικίνδυνε και δεύτερον ότι χρειαζόμαστε τον ΝΑΤΟ για να μα ε, υπερασπίσει από τέτοιε επιθέσει. Δεύτερη ερώτηση η στρατιωτικό αρχηγείο του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν εξέδωσε νέες οδηγίες για την υπογραφή συμβάσεων ώστε να, με οδηγίες για το πώς πρέπει να δαπανούν οι αρχηγοί 14 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ο στρατηγός Πετρέου στο υπόμνηνά του λέει ότι έχουμε ε, δαπανίσει πολλά ε, κεφάλαια συμβάσεων γρήγορα ώστε να καταπολεμούμε ώστε να με γεγονός να υπονομεύονται οι προσπάθειές μας στο Αφγανιστάν. Από τον περασμένο Ιούλιο σας διάβασα τον κείμενο το οποίο έχει υπογραφεί από μένα και άλλους 19 ε, βουλευτές που παραδόθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής και εκτιμώ το γεγονός ότι, ότι αντέδρασε άμεσα το ΝΑΤΟ και η ερώτησή μου είναι αυτό οφείλεται στην παρέμβασή σας, εφόσον μας είπατε ότι δεν γνωρίζετε το πρόβλημα, αλλά θα κάνετε κάθε τι το δυνατό για να παρέμβετε ή πρόκειται για απλή σύμπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Γενική Γραμματέα, ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Δύο παρατηρήσεις, τρει τρεις, Η επέκταση τη ανάλυση του πεδίου τη ε, απειλή με αποτέλεσμα το ΝΑΤΟ να είναι πλέον παρόν και να παρεμβαίνει στο σύνολο των, προβλημάτων που προκύπτουν σε πολιτικό επίπεδο. αναφερθήκαμε στις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, την κλιματική αλλαγή, την επιστημική ασφάλεια. Αυτό είναι ένα παράδοξο με αποτέλεσμα ένα οργανισμό άμυνα και ασφάλεια ξαφνικά να αρχίσει να ασχολείται με το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε πολιτικό επίπεδο. Δεύτερη παρατήρηση, αναφερθήκατε σε μια προληπτική παρέμβαση. Με, τι νομιμότητα, με τι νομιμότητα σε διεθνέ επίπεδο, στο πλαίσιο μια προληπτική ε, παρέμβαση από πλευρά ΝΑΤΟ τι ε, θα δίνει, ε, πώς νομιμοποιείται αυτή η παρέμβαση του ΝΑΤΟ. Και τρίτο παρατήρηση και ερώτηση αναφορθεί στις εξωτερικές σχέσεις. Παράλληλα βεβαίως με τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή πλαισιώνεται με πολύ αποφασιστικό τρόπο με ένα πλήρες σύστημα εξωτερικής εκπροσώπησης. Πώς φαντάζεστε το ρόλο του ΝΑΤΟ και των σχέσεων μεταξύ νατο και ευρωπαϊκής ένωσης τη στιγμή που η ευρωπαϊκή ένωση πλαισιώνεται όπως είπα με αυτό το σύστημα, αυτή την οργάνωση εξωτερικών σχέσεων. Ένα σύστημα που της έχει ανατεθεί από τη συνθήκη της Λισαβόνας και που περιλαμβάνει και τον τομέα της άμυνας. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις που ελπίζω θα μπορέσετε να δώσετε σε αυτά τα ερωτήματα κυρία Γενική Γραμματέα. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαού. Το λόγο έχει ο κύριος Κέλλαν για δύο λεπτά. Κύριε Γενική Γραμματέα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σαφή σας σχόλια ως προς τις ανάγκες μας. Ορισμένοι συνάδελφοι αναφερθήκαν στις ε, επιθέσεις στο κυβερνοχώρο. Σε περίπτωση μιας τέτοια επίθεσης μπορεί να υπάρξει κοινή ανταπάντηση όπως ισχύει στην περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης. Επίσης μπορούμε να έχουμε μια κοινή στρατηγική κατά των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο γιατί ξέρουμε ότι χρειάζονται χιλιοστά του δευτερολέπτου για να απαντήσουμε σε μια τέτοια επίθεση. Επίσης, μιλήσαμε για τις ε, υπηρεσίες πληροφοριών και πώς μπορούν να συνεργαστούν στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Μπορείτε να μας πείτε πώς προδεύει αυτή η ενδεχόμενη συνεργασία. Μιλήσατε για το συμπληρωματικό χαρακτήρα δράσης και συνεργασίας μεταξύ μελών του ΝΑΤΟ που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που δεν είναι. Και νομίζω ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τι θα γίνει με τις χώρες κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Μπορούν να συμμετέχουν σε κοινέ συνεδριάσεις. Ευχαριστούμε τον κύριο Κέλλεν. Η κυρία Λέζιν για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ράσμουσεν, και εγώ χαίρομαι που έχω την ευκαιρία σήμερα να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Σε δύο σημεία που αναφέρατε και εσείς ο ίδιος. προσπαθώ εδώ και καιρό να καταλάβω το περιεχόμενο μερικών συστάσεων της Ευρωπαϊκής ε, Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Μάλιστα να τις βρω και όλες τις συστάσεις αυτές στις 20 Φεβρουαρίου του 2010. Στις 16 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο στα συμπεράσματά του αναθέτει στην κυρία Άστο να καταρτήσει κατάλογο για ενίσχυση της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Στα συμπεράσματα τονίζει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ε, σύμφωνα με κάποιες συστάσεις που ήδη από το Φεβρουάριο του 2010 φέρεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει παραδώσει στον ΝΑΤΟ. Τι συστάσεις είναι αυτές, δεν τις γνωρίζω. Είναι δημόσιες και αν όχι γιατί. Και έχω και μία δεύτερη ερώτηση που αφορά τα όπλα μαζικής καταστροφής, το αναφέρετε και εσείς ο ίδιος ως προς τη στάθμευση πυρηνικών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο υπουργό ε, Εξωτερικών της Γερμανίας επιθυμεί απόσυρση, ενώ οι ΗΠΑ επιμένουν να παραμείνουν αυτά τα θαυμεμένα. Στην έκθεση που αναθέσατε για το 2020, να το 2020, Υπάρχει πρόταση αυτή η απόφαση να δεσμεύεται από μια συνενετική απόφαση της συμμαχίας. Εσείς τι λέτε, δεν θα πρέπει κάθε χώρα να ορίζει μόνη της εάν θα φιλοξενεί στην επικράτειά της πυρηνικά όπλα ή όχι. Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Λέζινγκ, ο κύριος Νέιτς, η κυρία Νέιτς, συγγνώμη, για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Είναι μεγάλη μας χαρά που βρίσκεστε μεταξύ μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν για άλλη μία φορά στο Κοινοβούλιο και σε αυτή την ε, διακοινοβουλευτική συνέλευση. Μας ε, σκιαγραφίσατε τη νέα στρατηγική κατά πάσα πιθανότητα του ΝΑΤΟ. Από τη μία πλευρά κατανοώ ότι θα επιμείνετε στην ανάπτυξη πολιτικών ικανοτήτων, αλλά εκεί που η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη προσπαθούν να αναπτύξουν αυτές τις πολιτικές ικανότητες για να ανταποκριθούν στις δικές τους δεσμεύσεις, στον τομέα της ε, πολιτικής ε, συνεργασίας θα ήθελα να σας τονίσω ότι δεν θα πρέπει να επικαλύπτονται οι προσπάθειες. Ως προς σχέση με τη Ρωσία, πολλοί προλαλήσαντες έμεσα ή άμεσα αναφέρθηκαν τις ε, δύσκολες σχέσεις γειτονίας, ιδιαίτερα όταν είναι γείτονες χώρες με τη Ρωσία. Άρα οι σχέσεις Ρωσίας-ΝΑΤΟ είναι κρίσιμες. Πώς ε, προβλέπετε να αναπτυχθούν στο μέλλον. Ευχαριστούμε την κυρία Νέιτς. Ο κύριος Τάνοκ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε για άλλη μια φορά εδώ στο Κοινοβούλιο, κύριε Γενικέ. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε καλύτερες ε, σχέσεις και να καταπολεμήσουμε τις επικαλύψεις. Εγώ ε, είμαι ε, αντιπρόεδρος της Διεπιτροπής με τις σχέσεις, ως προς σχέσεις με το ΝΑΤΟ και θα ήθελα να υποβάλω μία ε, διητή ερώτηση. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το βέτο της Τουρκίας σε σχέση με την ΕΠΑ ως προς την εκκρεμούσα κατάσταση στην Κύπρο και πώς μπορούμε να προωθήσουμε την ειρήνευση και την επανένωση της νήσου. Επίσης, πώς μπορούμε να διευρύνουμε ε, τη, τη σχέση μας με το ΝΑΤΟ. Όπως ξέρετε η Αλβανία είναι μέλος του ΝΑΤΟ αλλά δεν έχει ούτε καν ελεύθερες θεωρήσεις. Δηλαδή δεν έχει απαλλαγή από τις θεωρήσεις ενώ η Σερβία έχει ε, απελευθερωθεί από το καθεστώς των θεωρήσεων ενώ δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Πώς ε, το εξηγείτε αυτό. Και ως προς το κέρας της Αφρικής υπάρχει κοινή επιχείρηση η Αταλάντη και μία ξεχωριστή ε, επιχείρηση από πλευράς ΕΠΑ. Νομίζω ότι μη ε, συνδεδεμένες χώρες, οι αδέσμευτες χώρες, ε, δρούν σε αυτή την περιοχή. Αυτό αφορά αδέσμευτες χώρες όπως την Ινδία. Και η Ουκρανία επίσης θεωρεί ότι θα πρέπει να προωθήσει το θέμα της ε, προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μελλοντικά. Πώς βλέπετε το θέμα των επιθέσεων του κυβερνοχώρου σε σχέση με την ενδεχόμενη διεύρυνση του ΝΑΤΟ και των μελών του. Ο κύριος Σούλτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Γενικέ ε, Γραμματέα, για τη σύντομη παρουσίαση του νέου στρατηγικού δόγματος ε, και τους πέντε τομείς που αναφέρατε. Μιλήσετε για στρατηγική εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ σιγά σιγά μας έχει οδηγήσει σε σύγχυση γιατί έχει πολλές στρατηγικές εταιρικέ σχέσεις η Ένωση με τη Λευκορωσία, ξέρω εγώ, με την Ουκρανία, με τη Ρωσία διαπραγματευόμαστε και στρατηγική εταιρική σχέση με την Τουρκία ακούγεται κρεμή. Δεν Έχουμε συμμαχία ασφαλείας τώρα με 21 κράτη-μέλη που πάνω κάτω έχουν ατλαντικούς εταίρους. Και αν πρόκειται για στρατηγική εταιρική σχέση, πώς αξιολογείται τη δυνατότητα σύναψης εταιρικής σχέσης στρατηγικής και με τη Ρωσία. Ο πρώην Υπουργό Αμήνης Γερμανίας Φόλκερ Ρούε πρότεινε να μπει η Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. και από τον πρόεδρο Μετβέντεφ, το Think Tank και, το, και κάποιες άλλες δεξαμενές σκέψεις, το συζητούν και άλλοι και Γερμανοί και σοβαρά. Εσείς με τη νέα σας στρατηγική είστε προετοιμασμένοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Διεύρυνση προς Ανατολάς στην κυριολεξία του ΝΑΤΟ προβλέπεται, παίζει ρόλο στο νέο δόγμα. Κάποιοι συνάδελφοι το ανέφεραν ήδη και θέλω να το θέσω εγώ σαφέστερα τι λέτε για την πρόταση του Μετσβέτσεφ για μια νέα αρχιτεκτονική ασφαλεία στην Ευρώπη και πώς αξιολογείται τη δυνατότητα προσχώρησης της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ κύριος Λαντσπέργης για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ, σας ευχαριστώ και για την παρουσία σας και για την προθυμία σας να συνεργάζεστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη συμμετοχή της ε, Ρωσίας και τα όσα συζητήθηκαν από την εποχή που ανέλαβε ο κύριος Ομπάμα. Γίνονται μεγάλες συνομιλίες, που ακούγονται λόγια για ε, τις συμφωνίες συνεργασίας και ειρήνευσης και κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βάσει της δικής σας προσωπικής εμπειρίας και συμπεριφοράς υπάρχει καμιά ε, πιθανότητα να πείσετε τη Ρωσία ότι πάκτα σουν σερβάντα και όταν δεσμεύεσαι για κάτι και υπογράφεις θα πρέπει να το τηρείς και όχι να το ε, περιφρονής. Γιατί έτσι θα είναι η Ρωσία πραγματικός εταίρος. Βλέπε αξιόπιστος. Διαφορετικό από τη σημερινή κατάσταση συγκεκριμένη. Γιατί όταν το ΝΑΤΟ συνεργάζεται με κάποιον εταίρο, ενδεχομένως και μέλος του, θα πρέπει ο άλλος να είναι αξιόπιστος. Ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση ούτε καν έχουν αυτή την πρόθεση κάποια στιγμή να αξιοπιστεί. Βλέπετε τι έγινε πρόσφατα στον Κάφκασο. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκόμε, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματέα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά, αν πιστεύετε ότι η αναθεώρηση της στρατηγικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ αλλάζει σε ό,τι αφορά το δόγμα για τα μέσα μαζικής καταστροφής και τα πυρηνικά όπλα και την πυρηνική δύναμη συγκεκριμένα με βάση τη νέα φιλοσοφία που προωθεί η κυβέρνηση Ομπάμα στην ομιλία στην Πράχα και στην πρόσφατη διάσκεψη και θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Πιστεύετε το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ περιλαμβάνει, προβλέπει μια αντίδραση σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Καλύπτει την αντίδραση σε τέτοιου είδους επιθέσεις και πιστεύετε ότι ε, δεδομένης αυτής της νέας προσέγγισης που αφορά την πρόληψη κρίσεων και συνεργασία με αντίστοιχου οργανισμούς η στρατιωτική συμμαχία αλλάζει σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Και τέλος, εσεί ο Γενικό Γραμματέας του ΝΑΤΟ μπορείτε να πείτε στι Ηνωμένε Πολιτείε ότι η χρήση drones για επιλεκτικέ επιθέσει στο Αφγανιστάν δεν είναι αντίθετη στο διεθνές δίκαιο αλλά και αντιπαραγωγική σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα θύματα που προκαλεί και αποτελεί και ότι αυτό δεν είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και ότι θα πρέπει να σταματήσει γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί από τον κύριο Βάικολ για δύο λεπτά. Eh, Κύριε Γενική Γραμματέα, αυτά που μας είπατε για τις νέες απειλές προσέλκυσαν ε, πολύ το ενδιαφέρον μας. Πιστεύω όμως, όπως, και, όπως και πολλοί άλλοι, ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να δείξει να επιδείξει αυτό έλεγχο όταν μιλάμε για την, ε, τον εντοπισμό νέων απειλών. Απειλές που εμφανίζονται στο, στις φτωχές χώρες του κόσμου. Χώρες όπου υπάρχουν πολιτιστικές και θρησκευτικές διαφορές. Και θα ήθελα να θυμίσω ότι και εσείς συμβάλλατε σε αυτές τις παρανοήσεις και τις παρεξηγήσεις διότι είχατε μια συγκεκριμένη άποψη για τις γελιογραφίες που δημοσιεύθηκαν στις ε, δανεικές εφημερίδες στις δανέζικες εφημερίδες. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να σέβεται τη δημιουργικότητα, αλλά να παραμείνει ένας οργανισμός άμυνας, αποφεύγοντας τον κίνδυνο να θεωρηθεί ως, ως ε, αστυνομικός, παγκόσμιος, οικουμενικός αστυνομικός. Και υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος, τον οποίο αναφερθήκατε σήμερα την ιδέα μιας παγκόσμιας πυρηνικής, αντιπυρηνικής ασπίδας. Κάτι που δεν έγινε ποτέ δεκτό σαν μια λύση που προσφέρεται, που παρέχεται από τον ΝΑΤΟ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να δώσουμε την προτεραιότητα στις πολιτικές αποφάσεις. Και τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Μπορείτε να φανταστείτε τον ΝΑΤΟ να αναλαμβάνει έναν επικοδομητικό ρόλο στην αναζήτηση μιας ειρηνικής επίλυσης ή προωθώντας μια ε, ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, διότι εκεί βρίσκονται οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι και απειλές. Ευχαριστώ κύριε ε, Βάικελ. Με μεγάλη προσοχή παρατήρησα ότι σημείωνε τα όσα λέγατε ο Γενικός Γραμματέας και ε, ελπίζω να είναι εξίσου ακριβής και μεθοδικός και στην απάντησή του και τον ακούμε αμέσως. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις ε, και πολύ εύστοχες. Ζητώ συγγνώμη ε, εξ αρχής γιατί είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σύντομα αν θέλουμε να τελειώσουμε εγκαίρως. Πρώτος τον κύριο Ντονζόν για τη πολιτική, τις πολιτικές ικανότητες, μη στρατιωτικές και άλλοι το θέσατε. Ε, μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι τώρα μας απασχολεί αυτό, να δούμε πώς μπορούμε μέσα στο ΝΑΤΟ να δημιουργήσουμε μια μικρή πολιτική δομή ικανότητα, όχι ικανότητα να επεμβαίνει ε, σε πολιτικές δραστηριότητες στο ΝΑΤΟ το ίδιο, αλλά μια δυνατότητα να είμαστε σε καλύτερη θέση να συνεργαζόμαστε με άλλες οργανώσεις και άλλους οργανισμούς τύπου Ηνωμένων Εθνών, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμιας Τράπεζας, ε, την Τράπεζα για την Ανάπτυξη στην Ασία και άλλους φορείς που μπορούν να συνεισφέρουν ε, ε, στην πολιτική ανοικοδόμηση και στην ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη. Αυτό είναι μεταξύ άλλων ένα δίδαγμα του Αφγανιστάν αλλά και του Κοσφοπεδίου ότι αυτό που χρειάζεται είναι να βελτιώσουμε τη δυνατότητα που έχουμε να συνεργαζόμαστε με πολιτικές δομές, με πολιτικούς οργανισμούς και όχι στρατιωτικούς δηλαδή. Αυτό δεν έρχεται σε αντίφαση με ε, μεταρρύθμιση των δομών του ΝΑΤΟ. Σε καμία περίπτωση το αντίθετο. Προτεραιότητες θέτουμε. Ε, όπου χρειάζεται ε, αυξάνουμε τους μυς, μειώνουμε το λίπος, ε, τις περιττές δομές και ενισχύουμε τη συνεργασία μεταξύ των στρατιωτικών επιχειρήσεων και της πολιτικής ανάπτυξης. Το ΝΑΤΟ δεν θα είναι ποτέ πρωταγωνιστής της πολιτικής ανάπτυξης, αλλά θέλουμε να συνεργαζόμαστε καλύτερα με άλλους οργανισμούς. Ο κύριος Ντονζό με ρώτησε και για την Τουρκία. Εγώ δεν θεωρώ ότι ενδίδουμε ούτε στον ένα ούτε στον άλλον. Θεωρώ ότι είναι κοινή λογική να αναζητήσουμε ρεαλιστικούς τρόπους για να βελτιώσουμε τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Και πρότεινα ένα ρεαλιστικό δρόμο που δεν θίγει το ευαίσθητο θέμα της επίσημης αναγνώρισης της ε, Κυπριακής Δημοκρατίας, ούτε τις ε, διαπραγματεύσεις προνταξιακές Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αλλά ανάμεσα σε αυτά τα δύο θα πρέπει να βρούμε ρεαλιστικούς τρόπους να προχωρήσουμε. Και ανακεφαλαιώνω γιατί απαντώ και σε κάποιες άλλες ερωτήσεις που έγιναν σήμερα. Είναι πακέτο. Και ένα τμήμα του πακέτου είναι ότι όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα 27 θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Αλλά σε αντάλλαγμα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κινηθεί ε, και να εξυπηρετήσει κάποιες επιθυμίες που εκφράζουν μέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ ανέφερα τη Συμφωνία Ασφαλείας μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ανέφερα μια διευθέτηση ε, Τουρκίας και Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης η συμμετοχή μη κοινοτικών κρατών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων ε, για επιχειρήσεις ε, ενός τύπου Βοσνίας. Κατά τα άλλα, η Τουρκία είναι ο υπαριθμόν δύο χρηματοδότης της Ευρωπαϊκής Αποστολής στη Βοσνία, χωρίς να παίρνει μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Εμείς έχουμε στο Αφγανιστάν 19 ε, χώρες στην ISAF που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. 19 που δεν συμμετέχουν στις συνεδριάσεις μας. Βέβαια, σε τελική ανάλυση ε, την απόφαση την παίρνει το Συμβούλιο του Βορειοατλαντικό και για την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει το αντίστοιχο σε ό,τι την αφορά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν μη μέλη μας σε αυτή ε, τη διαδικασία. Και εφόσον συνεισφέρουν ε, και είναι αποκλεισμένοι από τη λήψη των αποφάσεων, κάτι πρέπει να γίνει. Και ελπίζω να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Κύριε Σουκάσκι, νομίζω ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρξει ένα συντονισμό Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για το Αφγανιστάν. Και επιτόπου στην Καμπούλ. Έχουμε ειδικού απεσταλμένου και χαίρομαι πάρα πολύ που διόρισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον ε, το δικό τη, που συνεργάζονται στενά με την πολιτική εκπροσώπηση του ΝΑΤΟ αλλά και τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών. Συνεργάζονται όλοι μαζί λοιπόν αγαστά και με την ISAF, τη Συμμαχία. Και γνωρίζονται. Είναι πραγματικά μια dream team στην Καμπούλα αυτή τη στιγμή. Στη Σύνοδο Κορυφή της Λισαβόνας επίσης θα υπάρξει μια συνεδρίαση όπου θα καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει σε μια Σύνοδο Κορυφή της ISAF. Έχω προσκαλέσει εκεί τον πρόεδρο Φαν Ρόμπεϊ και τον πρόεδρο Μπαρόσο να συμμετέχουν στη συνεδρίαση της ISAF στη Λισαβόνα όταν θα συζητήσουμε για το Αφγανιστάν. Λοιπόν, νομίζω ότι κάνουμε πολλά. Ακόμα προ τον κύριο Σουκάσκι που ζήτησε να συμμετέχει περισσότερο η Ρωσία στην αποστολή μας στο Αφγανιστάν. Το Δεκέμβριο μετέβη στη ε, Ρωσία και ζήτησα να στείλει ελικόπτερα στον Αφγανικό στρατό η Ρωσία. Και ε, αυτό τον καιρό το συζητούμε σε συνεργασία με τη Ρωσία. Έκαναν μια πρόταση και εκείνη και τη μελετούμε και ελπίζω να υπάρξει πρόοδος και εκεί. Κατά τα άλλα η Ρωσία ήδη ε, ε, μας δίνει διευκολύνσεις ε, διέλευσης για τα στρατεύματά μας προς το Αφγανιστάν. Επίσης συνεργαζόμαστε για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην Κεντρική Ασία και το Αφγανιστάν. Κύριε Λίσεκ, είχα μια συνάντηση με τον κύριο Γιανουκόβιτς τον Ουκρανό πρόεδρο, την περασμένη εβδομάδα. Σέβομαι πλήρως την απόφαση που έλαβε η νέα Ουκρανική κυβέρνηση ως προς τις σχέσεις της με το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει όμως να τονίσω ότι η αφετηρία του ΝΑΤΟ είναι η απόφαση που ελήφθη στη Σύνοδο Κορυφής του Βουκουριστίου το 2008, όπου είπαμε ότι και η Ουκρανία και η Γεωργία θα γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ, σε περίπτωση που το επιθυμούν και πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Προφανώς οι ίδιες θα αποφασίσουν πότε θα υποβάλουν επίσημη αίτηση ένταξης. Το ΝΑΤΟ είναι μια εθελοντική Ευρωπαϊκή ε, Συμμαχία. Σέβομαι πλήρως τις αποφάσεις των Ουκρανών, οι οποίοι είπαν και ότι θα τηρήσουν και τη δέσμευσή τους στο σημερινό πλαίσιο συνεργασίας που γίνεται ε, σε μια ειδική επιτροπή Ευρωπαϊκή, ε, ΝΑΤΟ ε, Ουκρανίας. Κύριε Ζιγκέρης, ζητήσατε πιο ορατή, προβεβλημένη παρουσία ε, του ΝΑΤΟ σε όλα τα μέλη του. Θα είναι ε, σημαντικό στοιχείο και του νέου στρατηγικού μας δόγματος και αυτό. Έχουμε την πρόθεση να φαινόμαστε περισσότερο, να είμαστε πιο ιρατοί και πιο προβεβλημένοι σε όλη την επικράτεια των ε, συμμάχων μας. Τι σημαίνει αυτό. Ασκήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα και επίση ε, επιτρέψτε μου να θυμίσω εδώ ότι οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ σήμερα στη Βαλτική επιβλέπουν τον εναέριο χώρο ε, εκ περιτροπής. Και είναι και αυτό παρουσία ορατή και απόδειξη αλληλεγγύης προς ε, τα μέλη της συμμαχίας μας. Η κυρία Κοπά επίσης αναφέρθηκε στην πολιτική ικανότητα, απάντησα ήδη σε αυτό νομίζω, ότι δεν θα υπάρξουν επικαλύψεις. Είναι ικανότητα βελτίωσης των σχέσεων της συνεργασίας μας με πολιτικούς οργανισμούς που πάντα θα έχουν εκείνο τον τελευταίο λόγο για την πολιτική ανάπτυξη. Κύριε Νεοφίτου. Συμφωνώ απολύτως με την ομάδα πυρογνωμόνων ότι η συνεργασία ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γίνεται με βάση την αμοιβαία διαφάνεια. Μα ήδη το τόνισα αυτό, άλλωστε. Συνεργασία μεταξύ των δύο οργανισμών θα σημάνει συνεργασία μεταξύ όλων των μελών και των δύο οργανισμών. Κυρία Γιαννάκου. Ποιε είναι οι πραγματικέ απειλές, ρωτάτε, στο σημερινό κόσμο. Δεν είναι συμβατικές, νομίζω. Δεν είναι οι πιο πιθανές οι συμβατικές. Σήμερα πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε νέες απειλές, όπως είναι η τρομοκρατία, οι πυραυλικέ επιθέσεις και θα μπορούσα να αναφέρω και χώρα. Το Ιράν. Έχει στη διάθεσή του πυράβλους βεληνικούς αρκετού για, να πλήξει στόχους στην Ευρώπη. Είναι πραγματική η απειλή αυτή. Τρομοκρατία, απειλές και ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αυτό δεν είναι θεωρητικό. Είδαμε την Εστονία πώς επλήγει πριν από λίγα χρόνια μες του διαδικτύου. Αυτές είναι οι νέες απειλές και οι νέες προκλήσεις. Και εμείς προτιθέμεθα να βελτιώσουμε τη δυνατότητα αντιμετώπιση τους. Ο κ. Σαρλάκη με ρώτησε γιατί να ασχολείται το ΝΑΤΟ δηλαδή με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Ε, οφείλω να σας πω ότι το ΝΑΤΟ οφείλει να ασχολείται με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, διότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο συνιστούν και πραγματική απειλή για τις στρατιωτικές μας δυνατότητες, αλλά και για όλη την κοινωνία. Και το ΝΑΤΟ έχει στη διάθεσή του ε, σχεδιασμό επιμελητεία, ε, δομές διοίκησης που να επιτρέπουν ένα πολύ αποτελεσματικό πλαίσιο αντιμετώπιση των επιθέσεων στον χώρο, αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούμε και στο μέλλον περισσότερο προς την κατεύθυνση αυτή. Τούτου λεχθέντος, είναι και ένας τομέας που θα μπορούσαμε να ευεργετηθούμε από στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Γιαννάκου με ρώτησε επίσης κάτι για το αν θα φύγει ποτέ το ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν. Η σύντομη απάντηση είναι βεβαίω, απολύτω. Το θέμα είναι πότε. Αλλά στόχος μας είναι να παραδώσουμε ε, στους Αφγανούς την ε, διακυβέρνηση της χώρας σε μια σταδιακή ε, μεταπατική περίοδο που ελπίζω να ξεκινήσει του χρόνου και να ενισχυθεί και να υλοποιηθεί ε, και η φιλοδοξία του κυρίου Καρζάη ότι θα είναι σε θέση μέχρι τα τέλη του 2014 να το πράξουν. Εγώ αναμένω τα διεθνή στρατεύματα να παραμείνουν και επέκεινα αυτή τη ε, ημερομηνία με ρόλο υποστηρικτικό. Αυτή τη στιγμή που οι Αφγανοί θα έχουν αναλάβει εκείνη τη διακυβέρνηση τη χώρα. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να είναι κυρίαρχοι στη χώρα τους ε, μια διαδικασία που να μην βασίζεται σε χρονοδιάγραμμα, αλλά σε διαδικασίε. Δεν μπορώ να σα δώσω ημερομηνία, αλλά η απάντησή σας είναι, ε, στην ερώτησή σα είναι καταφατική. Βεβαίω και θα φύγει το ΝΑΤΟ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκε. Ο κύριο Μαού με ρώτησε για προληπτικά μέτρα και ποια είναι η νομιμότητα και αν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι το ΝΑΤΟ πάντα θα δρά σε πλήρη συμφωνία με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές ε, του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. και η αποστολή μας στο Αφγανιστά ε, βασίζεται σε εντολή του ΟΗΕ όπως και η αποστολή μας στο Κωσυφοπαίδιο σε εντολή του ΟΗΕ και έτσι λειτουργούμε άλλωστε. Η μελλοντική διαχείριση κρίσεων θα βασίζεται πάντα ε, στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές ε, του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Εκτιμώ ε, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα δημιουργεί και συγκροτεί υπηρεσία εξωτερικής δράσης και έχω καλές σχέσεις συνεργασίας με την ύπατη εκπρόσωπο κυρία Άστον, όπως και με άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ συνεργάζομαι με όλα τα όργανα και με τον πρόεδρο Φαν και με τον πρόεδρο Μπαρόσο και με τον πρόεδρο Μπούσε, την κυρία Άστον βεβαίως και ε, είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ευκαιρία που έχω ε, να συζητώ σήμερα με βουλευτές. Νομίζω ότι σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συνεργαζόμαστε. Κύριε Κέλαμ. Ναι, για τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τώρα ε, αναπτύσσουμε αυτές τις δυνατότητες απόκρισης από κοινού, αν χρειαστεί. Είναι ένα νέο πεδίο και θα πρέπει πραγματικά να αναπτύξουμε τις δυνατότητες που έχουμε και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ως οργανισμός καθημερινά δέχεται επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, βελτιώσουμε την κοινή μας άμυνα εκεί. Κυρία Λόζενγκ, καλή ερώτηση για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σημειώσετε επίσης ότι γίνεται αναφορά σε κάποιες προτάσεις ή συστάσεις που ε, υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ΝΑΤΟ Δεν γνωρίζω εάν η ευρωπαϊκή πλευρά της έχει δημοσιεύσει, γιατί εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημοσιεύσει. Επιβεβαιώνω όμως ότι έχω λάβει συγκεκριμένες προτάσεις. Και θα ήθελα να σα επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ορίζουν ρητά ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις προτάσεις και το τονίζω με ικανοποιούν οι προτάσεις που λάβαμε, αλλά δεν νομίζω ότι δίνουν την απαραίτητη πλατφόρμα για μια πραγματική καμπή στις σχέσεις μας. Δηλαδή θα πρέπει να τις υπερβούμε και προσβλέπω στη συνάντηση που θα έχω με την υπατή εκπρόσωπο και με άλλα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πυρηνικά. Και βέβαια τελικά η πολιτική ασφαλείας και η πυρηνική είναι αποφάσεις εθνικές. Ωστόσο, έχουμε συμφωνήσει στο ΝΑΤΟ ότι αποφάσεις που λαμβάνονται σε μία χώρα μπορεί να έχουν ε, επιπτώσεις σε αποφάσεις άλλων χωρών. Γι' αυτό δεσμευτήκαμε να έχουμε διαβουλεύσεις πριν, παίρνουμε, πριν πάρουμε αποφάσεις και πριν κάνουμε κάποια βήματα. Δηλαδή να υπάρχει ένα πνεύμα συνενετικό στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Και βέβαια τονίζω ότι τέτοιου είδους αποφάσεις τελικά είναι θέματα εθνικών κυβερνήσεων, αλλά μπορεί και μια χώρα να αποφασίσει ότι για να αποφασίσει θα συνεργαστεί με τους άλλους. Ανεμινέιτς. Και ο κύριος Σούλτς με ρώτησαν για τη Ρωσία. Και πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις μας. Πολύ σημαντική ερώτηση. Πρώτον, ρωτάει ο κύριο Σούλς, θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη Ρωσία μελλοντικό μέλο του ΝΑΤΟ. Να σα πω. Ομολογώ ότι στο άρθρο 10 του Βορειοατλαντικού Συμφώνου ορίζεται ότι η συμμαχία μπορεί να καλέσει οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα που είναι σε θέση να συνεισφέρει στην ευρωατλαντική ασφάλεια και που είναι σε σχέση να ε, διαδώσει τις αρχές ε, της, του συμφώνου, μπορούμε να καλέσουμε μια τέτοια χώρα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αυτό ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε, υπό την έννοια αυτή δεν αποκλείουμε κανέναν. Βέβαια, τούτου λεχθέντος. Δεν νομίζω ότι είναι ρεαλιστική προοπτική να θεωρεί κανείς τη Ρωσία μέλος του ΝΑΤΟ. Πάντως δεν το έχουν ζητήσει. Και ο Ρώσος πρέσβης μάλιστα στο ΝΑΤΟ τόνισε ότι δεν ποτέ πρόκειται να ζητήσουν κάτι τέτοιο. Πάντως νομίζω ρεαλιστική προσέγγιση θα ήταν να αναπτύξουμε αυτό που θα ονόμαζα στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Διότι, παρά το γεγονός ότι έχουμε και τις διαφορές μας με τη Ρωσία και τις διαφωνίες μας για τη Γεωργία και για άλλα θέματα, υπάρχουν σαφέστατα τομείς όπου είναι κοινά τα συμφέροντα ασφαλείας μας. Κατά τα άλλα, το Αφγανιστάν είναι ένα μόνο αλλά και καταπολέμηση της τρομοκρατίας, των ναρκωτικών, της πειρατείας. Και σας είπα και την αντιπυραυλική ε, άμυνα ως ενδεχόμενο τομέα συνεργασίας επίσης. Και νομίζω ότι σε αυτούς τους τομείς θα πρέπει να αναπτυχθεί ε, συνεργασία, εκεί που έχουμε τις ίδιες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε και οι δύο. Και επιτρέψτε μου να τονίσω κάτι ακόμα. Στην αντιπυραυλική άμυνα όπως είπα ήδη, είναι πραγματική απειλή. Και απέναντι σε μια πραγματική απειλή χρειαζόμαστε πραγματική άμυνα. Εάν αποφασίσουμε να αναπτύξουμε ένα σύστημα αντιπυραυλικό του, του ΝΑΤΟ, έχει νόημα να καλέσουμε και τη Ρωσία να συνεργαστεί και στρατιωτικά. Διότι θα μας δώσουν διευκολύνσεις, καλύτερη κάλυψη, πιο αποτελεσματική και πολιτικά όμως, διότι θα αποδείξει ότι αυτή η αντιπυραυλική άμυνα δεν στρέφεται κατά της Ρωσίας. Αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πραγματικά μια στρατηγική ασφαλείας, ευρωατλαντική, που να καλύπτει ε, την Ευρώπη και τον Ατλαντικό από το Βανκούβερ μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Έτσι θα μπορούσαμε να μιλάμε για πραγματική ασφάλεια. Αυτό είναι εκείνο που έχει σημασία για τον κόσμο. Έτσι βλέπω εγώ τη σχέση μας με τη Ρωσία. Ο κύριος Τάνοκ με ρώτησε για τα Βαλκάνια. Το όραμά μου είναι όλες οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στην Ευρωατλαντική δομή στο ΝΑΤΟ δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα γίνει με διαφορετικές ταχύτητες. Συμφωνώ, πρέπει να σεβαστούμε διαφορές σε ό,τι αφορά τις προσδοκίες για προσχώρηση στους ευρωατλαντικές δομές αυτών των χωρών, αλλά έχουν σημειωθεί πρόοδοι. Έχουμε έχουμε ε, ε, ήδη συμφωνήσει κάτι με το Μαυροβούνιο και με τη Βοσνία. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τα Σκόπια διαδικασίες ένταξης μόλις βρεθεί στο θέμα της ονομασίας μια ικανοποιητική λύση και ελπίζω να υπάρξει και πρόοδο στις σχέσεις μας με τη Σερβία επίσης. Είμαι λοιπόν αισιόδοξο για τις μελλοντικέ εξελίξεις στα Βαλκάνια. Η κυρία Γκόμες με ρώτησε για την, τον νέο στρατηγικό σχεδιασμό. Διαπραγματευόμαστε αυτή τη στιγμή το νέο στρατηγικό σχεδιασμό με στόχο αφενός να προωθήσουμε το σημαντικό όραμα ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα, ενώ ταυτόχρονα λέμε ότι εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν πυρηνικά όπλα, χρειαζόμαστε και ένα αποτελεσματικό σύστημα αποτροπής. Πρέπει ωστόσο θα καταβάλουμε προσπάθειες για να περιορίσουμε την εξάρτηση από, το, από τα πυρηνικά όπλα. Το κυβερνοχώρος. Ίσως ενδεχομένως να καλύπτεται από το άρθρο 5 κάποια στιγμή. Με βάση το σύμφωνο τη συνθήκη, οποιοδήποτε σύμμαχος μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις εάν αισθάνεται ότι απειλείται δυνάμει του άρθρου 4 και αν οι διαβουλεύσεις καταλήξουν συμπέρασμα ότι πρέπει να ληφθούν, να γίνουν ενέργειες, τότε μπορεί να τεθεί σε ισχύ το άρθρο 5. Δυνητικά λοιπόν η απάντηση είναι ναι. Και τέλος ο κύριος Βάγκελ. Όχι, απαντώ. Δεν θα γίνει ο οικουμενικός αστυνομικός το ΝΑΤΟ. Ασφαλώς όχι αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους λαούς μας αποτελεσματικά στο σημερινό κόσμο, πρέπει παράλληλα να αντιμετωπίσουμε και να λάβουμε υπόψη μας με αποτελεσματικό τρόπο νέες απειλές όταν μιλάμε για τρομοκρατία και να καταπολεμήσουμε και να πολεμήσουμε στις ρίζες του στην τρομοκρατία όπως συμβαίνει στο Αφγανιστάν. Δεν θα παίξουμε λοιπόν ρόλο παγκόσμιου αστυνομικού, αλλά θα εξασφαλίσουμε την μια αποτελεσματική προστασία για τις χώρες και τους πολίτες τους. Και τέλος έρχομαι στο Μεσανατολικό. Είναι κάπως πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλάμε σε αυτό το στάδιο, σε αυτή τη φάση, για οποιοδήποτε ρόλο των ε, διεθνών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα ειρηνευτική συμφωνία. Αλλά αν ακολουθήσουμε τις, ας ακολουθήσουμε τις σας και ας είμαστε αισιόδοξοι και ας υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία. Τότε πιστεύω ότι θα χρειαστεί η παρουσία διεθνών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή που θα παρακολουθούν και θα ελέγχουν αυτή τη ειρηνευτική διαδικασία, αυτή τη συμφωνία. Μπορούμε να φανταστούμε ρόλο του ΝΑΤΟ σε αυτή την περίπτωση. Δεν το ξέρω. Η απάντησή μας μέχρι τώρα ήταν ότι αν υπάρξει συμφωνία ειρήνης, εάν ε, τα μέρη ζητήσουν τη βοήθειά μας και εάν τα Ηνωμένα Έθνη η εντολή ε, εξουσιοδοτήσουν μια τέτοια αποστολή, τότε οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟΥ θα είναι έτοιμοι να εξετάσουν αυτό το ενδεχόμενο. Αυτή είναι η στάση μας επί του παρόντος. Το πρώτο βήμα όμως θα είναι να υπάρξει μια συμφωνία ειρήνης και αυτή θα είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και εύχομαι στις ενδιαφερόμενες πλευρές κάθε επιτυχία διότι αυτή η σύραξη έχει δημιουργήσει έχει είναι αφορμή για πάρα πολλές εντάσεις και σειράξεις σε άλλες περιοχές του πλανήτη και οπωσδήποτε θα είναι πιο ειρηνικός ο κόσμος, ο πλανήτης μας, αν υπάρξει λύση σε αυτή τη διαφορά. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Νομίζω ότι ε, θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ορισμένα συμπερασματικά ε, σχόλια, ε, αν το επιθυμεί και ο κύριος Ντανζόν. Νομίζω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα σχόλια του κυρίου Λίζεκ, διότι συζήτησα το θέμα με τον πρόεδρο της Γεωργίας, ο οποίος βρέθηκε φευγαλέα στις Βρυξέλλες και ίσως ε, κύριε Γενικέ μπορείτε να μας πείτε ορισμένα, μπορείτε να σχολιάσετε την κατάσταση της Γεωργίας με βάση την πρόσφατη αυτή επίσκεψη στις Βρυξέλλες. Πράγματι, αναφέρθηκα στην Ουκρανία και ως προς τη Γεωργία η θέση μας είναι η ίδια, δηλαδή η απόφαση που λάβαμε στη διάσκεψη του Βουκουρεστίου το 2008 το ΝΑΤΟ αποφάσισε στο Βουκουρέστι το 2008 ότι η Γεωργία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θα γίνει μέλος υπό τον όρο ότι πληρούν τα αναγκαία κριτήρια. Και με βάση τα γεγονότα του Αυγούστου του 2008 προβήκαμε στη σύσταση μιας επιτροπής ΝΑΤΟ-Γεωργία και συνεργαζόμαστε με τη Γεωργία. Στα πλαίσια αυτής της Επιτροπής έχουμε συναντήσει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε πολιτικό επίπεδο. Η Γεωργία έχει βλέψεις προς την Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία και θα συνεχίσουμε να υποβοηθούμε τη Γεωργία για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, κοινωνικές ε, μεταρρυθμίσεις προς αυτή την κατεύθυνση την Παρασκευή αυτή την εβδομάδα θα παρευρεθώ στην Τυφλίδα και θα έχω μια πολιτική συνάντηση με τους ε, πολιτικούς αρχηγούς και αυτό είναι ένα άλλο βήμα που συνάδει προς τους, με τους απότερους στόχους μας. Δηλαδή, η συνεργασία με τη Γεωργία θα συνεχιστεί στα πλαίσια της διμερούς αυτής επιτροπής ΝΑΤΟ-Γεωργία. Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ και για αυτή την απάντηση όπως και για όλες τις άλλες που ήταν ιδιαίτερα ακριβείς ως προς το περιεχόμενο. Είχαμε μεγάλη ε, παρουσία, πολλά επιχειρήματα ακούστηκαν, πολλές παρεμβάσεις μέσα στα πλαίσια του χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι η σημερινή ε, συνεδρίαση ήταν ε, ιδιαίτερα επικοδομητική. Είδαμε ποιες είναι οι νέες ε, προκλήσεις που προβάλλονται και οι νέες δυνατότητες που διανοίγονται με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας και βεβαίως οι νέες σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Αλλά βεβαίως οι προσδοκίες έχουν πάντα ανθρώπινη διάσταση και αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρχει μία επικοινωνιακή πολιτική που υπάρχει μεταξύ ημών και ημών. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά θέματα εν εξελίξη αλλά νομίζω ότι οι συναντήσεις μας σε τακτά χρονικά διαστήματα βοηθούν την, τις όλες διαδικασίες συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Σας ευχαριστώ πολύ. πριν ε, ε, αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για τη συνεργασία και τους εύχομαι ε, καλή επιστροφή με τα προβλήματα που υπάρχουν βεβαίως στην εναέρια κυκλοφορία. Σας εύχομαι καλή επιστροφή παρά τα προβλήματα λοιπόν.